Καλημέρα σας, ε, συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας. Μετά τη χθεσινή παρουσίαση από την πλευρά του κυρίου εισηγητή και των συναδέλφων των εγγράφων εργασίας ε, για την ε, σε επιπτώσει ε, στην οικονομία τη νομοποίηση Παραδείγματος όταν μιλήσαμε για τράπεζες, για χρηματοοικονομικά. Σήμερα θα μπούμε σε ένα ειδικό θέμα που θα μας επιτρέψει να έχουμε περαιτέρω χρήσιμα στοιχεία για τις εργασίες μας. Το πρώτο κλάστερ εφέρει τον τίτλο αστυνόμευση βάση στρατηγικών πληροφοριών ε, ως προσέγγιση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τη διαφθορά και του ξεπλήματος νομικοσυμμετός. Θα ακούσουμε τον κύριο Φαρσίου που είναι διευθυντή τη δικαστικής αστυνομίας του Βελγίου που θα μιλήσει για τη χρήση των πληροφοριών από τη Βελγική αστυνομία, τον Τριού Χάρη, ο οποίο είναι υπαρχηγό ε, του τμήματο τη ε, αστυνομία τη Βόρεια Ιρλανδία, που θα μα μιλήσει για τι αστυνομικέ δράσει του Ηνωμένου Βασίλειου, τον κύριο Χούθ, ε, ο οποίο προέρχεται από την Βεσφαλία στη Γερμανία και θα μα μιλήσει για τη χρήση των πληροφοριών από την πλευρά τη ε, γερμανική εγκληματολογική αστυνομία και επίση την Τωρέα Αμίτσι, ε, η οποία είναι αρμόδια για την ε, αστυνομική συνεργασία και τις σχέσεις με την Κυριοπόλη και τη ΕΠΟΛ και θα μιλήσει για την ενδυνάμωση και την εφαρμογή του δικαίου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτησή μας θα διεξαχθεί ο συνήθως, 15 λεπτά θα έχει διαθέσει το κάθε ομιλητής και κατόπιν θα περάσουμε στη συζήτηση. Οι συνάδελφοι θα εκθέσουν τις σκέψεις τους και τις ερωτήσεις τους. Και πάλι θα ξαναδώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους. Έχετε λοιπόν 15 λεπτά, καταρχήν ο κύριος Φαρσή. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα το πρωί θα σας εξηγήσω και θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες για την προσέγγιση που ακολουθούμε στο Βέλγιο όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών που οδηγεί στην προσέγγιση των αστυνομικών αρχών και τι ρόλο παίζει στην καταπολέμηση του εγκλήματος γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα του οργανωμένου εγκλήματος. Η ανταλλαγή πληροφοριών λοιπόν είναι μια ευρία έννοια και ένας πολύ ευρύς τομέας δραστηριοτήτων. Για τον ε, ορισμό πρέπει να ξέρουμε ότι είναι άλλο πράγμα η πληροφορία απλώς και άλλο η ανταλλαγή πληροφοριών. Η πληροφορία απλώς είναι μια πληροφορία που έρχεται που δεν έχει τύχει καμία επεξεργασία. Ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών καλύπτει, είναι επεξεργασμένη και καλύπτει πάρα πολλού τομεί. Τον στρατιωτικό, τον οικονομικό, τον δημοσιονομικό και ε, βέβαια το έγκλημα, αυτό που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Η ανταλλαγή πληροφοριών λοιπόν γίνεται σε τρία επίπεδα. Είναι στρατηγικός ο χειρισμός, μπορεί να είναι χειρισμός τακτικής και μπορεί να είναι και επιχειρησιακό το επίπεδο επεξεργασίας της ανταλλαγής αυτής πληροφοριών. Είναι κάτι συγκεκριμένο και κάτι εικονικό και ε, συλλέγεται η πληροφορία και γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών από βέβαια ανθρώπους, από ανθρώπινους σπόρους, από ανοιχτές πηγές ε, που μπορεί να γίνεται ο χειρισμός αυτός ε, απόρριτα ή όχι. Πρέπει να ξέρουμε ότι στο Βέλγιο η αστυνομία εδώ και πολλά χρόνια έχει οθετήσει μία προσέγγιση που βασίζεται σε αυτό που λέμε intelligence-led policing. Δηλαδή είναι η δράση των αστυνομικών αρχών που βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και εκφράζει την βούληση να λειτουργεί η αστυνομία βάσει της ανταλλαγής πληροφοριών. Οι εγκληματικέ δραστηριότητε είναι διαφορετικού τύπου βέβαια και γι' αυτό η αστυνομία και τα δικαστήρια πρέπει να εγκαταλείψουν την στάση που είχαν μέχρι τώρα που ήταν να κάνουν τον πυροσβέστη, να τρέχουν δηλαδή πίσω από το έγκλημα για να σβήνουν τη φωτιά επειδή δεν την πρόλαβαν ή επειδή δεν μπόρεσαν να την ελέγξουν έγκαιρα η ανταλλαγή αυτή πληροφοριών για την οποία σας μιλάω σήμερα αποτελεί τον τρίτο δρόμο ανάμεσα στην καθημερινή δουλειά της αστυνομίας που είναι η αντίδραση στα γεγονότα δηλαδή και την τρέχουσα πρακτική που είναι η πρόληψη και η αποτροπή του εγκλήματος. Μια πρακτική που τελικά δεν έχει καταφέρει να ελέγξει το έγκλημα, το οργανωμένο. Μέσα στην αστυνομία για να πετύχουμε με την προσέγγιση μας αυτή πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται τόσο για μια τεχνική όσο για μια πραγματική φιλοσοφική διάσταση της αντιμετώπισης. Ξέρετε ότι όλοι οι καλοί μπάτς εντό αγωγικών τι κάνουν, ψάχνουν την σωστή πληροφορία, τον σωστό πληροφοριοδότη για να πετύχουν. Όμως βασίζονται πολύ στο ένστικτο και γι' αυτό και δεν είναι τόσο αποτελεσματική μακροπρόθεσμα. Η προσέγγιση που προσπαθούμε εμείς να αναπτύξουμε μέσα στην ε, Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου είναι μια προσέγγιση και πλήρης και συμπαγής. Είναι πλήρης γιατί λαμβάνει υπόψη τα τρία επίπεδα της ανταλλαγής πληροφοριών του στρατηγικού χαρακτήρα, της τακτικής και του επιχειρησιακού χαρακτήρα, όπως επίσης λαμβάνει υπόψη και τη σχέση μεταξύ τους. Η πρώτη το πρώτο επίπεδο, το στρατηγικό, βοηθά για να καταλάβουμε καλύτερα το πλαίσιο, για να έχουμε μια εικόνα των μορφών του εγκλήματος και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του σήμερα και του αύριο. Ε, συνεργαζόμαστε βέβαια και με άλλους φορείς, με την Interpol, την Europol, ακόμα και τον Ηνωμένα Έθνη. Και πρόκειται για ανταλλαγή πληροφοριών με πληροφορίες που στην αρχή μπορεί να φαίνονται εντελώ ανώδυνες, αλλά οι οποίες μας βοηθούν εφόσον αναλυθούν να σχηματίσουμε καλύτερα την εικόνα του εγκληματικού φαινομένου ή του εγκληματικού χώρου. Για παράδειγμα, <clears throat> πώς προμηθεύεται η Ευρώπη κοκαίνη ή πώς κυκλοφορούν στην Ευρώπη οι διάφορες αλβανικές μαφίες. Τώρα το δεύτερο επίπεδο τακτικής. Εδώ πέρα πρόκειται για, μια, για ένα σχεδιασμό δράσεων που έχουν ως στόχο την ε, εγκληματική δραστηριότητα, αλλά πολύ συγκεκριμένα στο χώρο και στο χρόνο. Σαν παράδειγμα θα σας δώσω, να αν ξέρουμε ας πούμε ότι σε ένα Δήμο ε, κλέβονται πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια βέβαια πουλούνται παράνομα. Ή αν υπάρχει κάποιο μαγαζί το οποίο ανήκει στον εγκληματικό χώρο της Νιγηρίας και ε, δουλεύουν εκεί οι κοπέλες συνοδοί που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπινων όντων. Αυτά είναι τακτικού χαρακτήρα. Και έχουμε τώρα στο επιχειρησιακό επίπεδο που έχει να κάνει με στοιχεία πολύ συγκεκριμένα πληροφοριών που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε έναν ύποπτο. Για παράδειγμα, αν βρούμε τον αριθμό του κινητού ενός ύποπτου ή τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ενός συνένοχου και μπορέσουμε και εντοπίσουμε στη συνέχεια το τηλέφωνο αυτό, δηλαδή μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε ή βρούμε το αυτοκίνητο ή αν βρούμε τη από κάποια ληστεία. Βέβαια αυτές οι τρεις μορφές είναι λέδετες μεταξύ τους. Δεν μπορούμε, αν δεν έχουμε το πλαίσιο, να προχωρήσουμε και δεν μπορούμε να σχηματίσουμε εικόνα για μια εγκληματική οργάνωση αν δεν αναλύσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και στα τρία επίπεδα. Αυτή λοιπόν η ε, πλήρης προσέγγιση λειτουργεί και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Όμω είπαμε ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι και συμπαγή. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις πλευρές, την αστυνομία, τι υπηρεσίε πληροφοριών, όλους τους φορείς. Γιατί είναι μια υπόθεση όλων. Είτε πρόκειται για τον αστυνόμο τη γειτονιά, είτε πρόκειται για τον ειδικό στι ενδείξει, είτε πρόκειται για τον ανακριτή, είτε πρόκειται για αυτόν που ψάχνει στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν η προσέγγιση αυτή είναι τόσο από πάνω προς τα κάτω, top down, όσο και από κάτω προς τα πάνω, bottom up. Η ανταλλαγή πληροφοριών στρατηγικού επίπεδου συνήθως πηγαίνει από πάνω στην ιεραρχία προς τα κάτω, ενώ ε, της τακτικής λειτουργεί μέσα σε ένα διάμεσο επίπεδο, γιατί γίνεται έρευνα και ξεκινούν έρευνες με συγκεκριμένους στόχους. Όταν φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο, αυτό συνήθως γίνεται από τους ανθρώπους που δουλεύουν επί τόπου, την αστυνομία δηλαδή που δουλεύει επί τόπου, αλλά φυσικά εδώ χρησιμοποιούνται και οι αναλυτές που αναλύουν τις διάφορες ενδείξεις. Πρόκειται δηλαδή για μια διτή προσέγγιση, top-down και bottom-up. Το πλεονέκτημά της είναι ότι προσφέρει μια καλύτερη εικόνα της ασφάλειας και της εγκληματικότητας αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε τώρα στην εικόνα της ασφάλειας. Σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο όμως δικαστικών διαμερισμάτων λειτουργεί αυτό στο Βέλγιο. Εμείς προτιμάμε να μιλάμε για, την, ε, για τον μόνιμο διαγνωστικό χαρακτήρα της ασφάλειας. Είναι δηλαδή μια προσέγγιση που σημαίνει ότι δεν μας φτάνει η εικόνα, η φωτογραφία της κατάστασης μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά θέλουμε να καταλήγουμε και σε συμπεράσματα για να υιοθετήσουμε μέτρα θεραπευτικού χαρακτήρα, για να χρησιμοποιήσω πάλι την ιατρική ορολογία. Στο Βέλγιο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο ασφάλειας που έχει αναπτύξει η αστυνομία και έχει εγκριθεί και από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Ε, πρόκειται για ένα σχέδιο με διάρκεια τέσσερα χρόνια που καθορίζει προτεραιότητες καταπολέμησης των εγκληματικών φαινομένων. Ε, πριν ορίσουμε το σχέδιο αυτό, οι υπηρεσίε της αστυνομίας σε συνεργασία με την δικαιοσύνη και τα Υπουργεία και τους ακαδημαϊκούς ανέπτυξαν αυτό που ονομάζουμε εθνική εικόνα της ασφάλειας, που βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα για το έγκλημα, ελαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς, την Europol για παράδειγμα, με την έκθεση ΣΟΚΤΑ, ε, στοιχεία από την Interpol, αλλά και από οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και μετά από συνομιλίες με καθηγητές, ε, ε, διευθυντές Υπουργείων κλπ. Αυτή η εικόνα λοιπόν μας βοηθάει πολύ να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό των δράσεών μας. Η εικόνα αυτή μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε βασικές κατευθυντήριες γραμμές, σε προσανατολισμούς δηλαδή. Τέθηκαν θέματα προθεσμιών. Ε, είπαμε κάποια στιγμή ότι η εικόνα αυτή δεν φτάνει για να αναπτύξουμε δραστηριότητες ε, επιτόπου ότι αυτή η εικόνα είναι μια φωτογραφία μια συγκεκριμένη στιγμή που ξεπερνέεται πάρα πολύ γρήγορα από τα γεγονότα. Ακριβώ επειδή ο εγκληματικό κόσμο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν λαμβάνει υπόψη ε, τα στοιχεία τακτική που μπορούν να μα βοηθήσουν καλύτερα να καθορίσουμε τι δράσει μα. Γι' αυτό και μιλήσαμε για τον μόνιμο διαγνωστικό χαρακτήρα της ε, ασφάλειας ανά διαμέρισμα. Και έτσι χρησιμοποιούμε και την εικόνα αλλά και τα στοιχεία που συλλέγονται σε καθημερινή βάση από την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Για να καταλήξουμε σε, σε μια πλήρη διάγνωση αλλά και για να καταδείξουμε καλύτερα ε, ποιε είναι οι εγκληματικέ οργανώσεις που δρούν ε, στον χώρο μας. Και γι' αυτό λάβαμε υπόψη μας τις εγκληματικέ ε, ροές, δηλαδή τα εγκληματικά φαινόμενα τα οποία βέβαια γνωρίζει και συμπεριλαμβάνει στις στατιστικές της η Εθνική Αστυνομία. Λαμβάνουμε υπόψη μας επίσης τους δράστες και τις ε, εγκληματικές οργανώσεις που ξέρουμε ότι δρούν στη χώρα και το δεύτερο, το τρίτο συγγνώμη που λαμβάνουμε υπόψη μας είναι τον εγκληματικό χώρο, δηλαδή γεωγραφικά που λαμβάνουν χώρα τα εγκληματικά φαινόμενα. Θελήσαμε λοιπόν, λαμβάνουμε υπόψη μας ε, του γεωγραφικό χώρο, βάσει των όσων έχει ορίσει ο Καναδός ο ερευνητής και εγκληματολόγος Μωρίς Κουσόν, ε, λάβαμε υπόψη μας λοιπόν την γεωγραφία που λαμβάνουν χώρα τα εγκλήματα ως χώρο δίωξης, αλλά λάβουμε επίσης υπόψη μας και που ζουν οι εγκληματίες και ποιοι είναι οι χώροι ψυχαγωγίας τους, δηλαδή πού συγκεντρώνονται και που οργανώνουν τα εγκλήματό τους. Είτε πρόκειται για μπάρ, είτε πρόκειται για άλλους χώρους, ε, παράνομου τζόγου κλπ. κλπ. Η μεθοδολογία λοιπόν της διάγνωσης αυτής μας επιτρέπει να έχουμε και την φωτογραφία όπως είπαμε πριν τη στιγμή της συγκεκριμένης του εγκλήματος αλλά έτσι μπορούμε να ελέγξουμε και τον περίγυρο των ε, εγκληματικών οργανώσεων βάσει αυτών των τριών παραγόντων που σας είπα πριν. Στο Βέλιο υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε τα σταυροδρόμια της πληροφόρησης στο Βέλιο. Εκεί γίνεται δηλαδή η ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία που έχουμε για το έγκλημα. Λαμβάνουμε υπόψη μας λοιπόν τα αστυνομικά δεδομένα από τα δεδομένα επίσης που έχουμε και από άλλες χώρες και έτσι μπορούμε να δώσουμε και εμείς πληροφορίες επιχειρησιακού χαρακτήρα σε καθημερινή βάση από την αστυνομία και να οργανώσουμε τις δράσεις μας καλύτερα. Έρχομαι πάλι στην προσέγγισή μας που σας είπα ότι είναι πλήρης και συμπαγής. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε και με την μόνιμη διάγνωση όσον αφορά την ασφάλεια στο Βέλγιο αλλά και την παρακολούθηση. Η ιδέα είναι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τη διάγνωση, αλλά στη συνέχεια να ανταποκρινόμαστε ακόμα καλύτερα στην πραγματικότητα. Και στα τρία επίπεδα, το στρατηγικό, το τακτικής και το επιχειρησιακό, προσπαθούμε να μειώσουμε τον χρόνο ανάμεσα στα γεγονότα και τις δράσεις μας. Σε διεθνές επίπεδο το Βέλγιο βοηθάει διεθνή όργανα όπως είναι την Europol και μπορούμε καλύτερα ακόμα να βοηθήσουμε σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν με την μέθοδο αυτή. Και έτσι αναλύουμε καλύτερα, λαμβάνοντα υπόψη μας την έκθεση ΣΟΚΤΑ, αλλά και ε, το AWF, που ονομάζεται Focal Points τελευταία, και βοηθούμε έτσι στα πλαίσια της European Policy Cycle. Ο τελικός στόχος μας λοιπόν είναι, σεβόμενοι το θεσμικό και το νομικό πλαίσιο, να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα και να προλαμβάνουμε το έγκλημα αναλύοντας τις πληροφορίες και ακολουθώντας μια μόνιμη πολιτική ε, που οδηγεί σε περισσότερες πληροφορίες. Δεν διαπιστώνουμε μόνο το έγκλημα, αλλά λαμβάνουμε υπόψη μας και ό,τι πληροφορίες έχουμε από το σύνολο των υπηρεσιών μας. Έτσι, οι πληροφορίες μας αυτές αποτελούνται και από διαπιστώσεις, αλλά και από πληροφορίες ε, γύρω από το έγκλημα. Εν κατακλείδη, η ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης της πύρους και συμπαγούς αποτελεί για τις υπηρεσίες μας κάτι πάρα πολύ θετικό και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της αστυνομίας και κάθε υπηρεσίας ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χάρης από τη Βόρεια Ιρλανδία, ο οποίος είναι υπαρχηγός του εγκληματολογικού για να μας μιλήσει για τη δική του εμπειρία σε σχέση με την αστυνόμευση βάση στρατηγικών πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Λέγομαι Ντρου και είμαι υπεύθυνο για τις εγκληματολογικές έρευνε στη Βορειοϊρλανδία και περιλαμβάνεται και το σοβαρό έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα, η παρακολούθηση βάση πληροφοριών και ανάλυση ε, των εγκληματολογικών θεσίων. Είμαστε ε, μια υπηρεσία που υπηρετεί 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους και η Βορειοϊρλανδία είναι πάρα πολύ ασφαλής περιοχή, αλλά έχουμε το μόνο σύνορο, με το είμαστε στο μόνο σύνορο του Ηνωμένου Βασιλείου, το Χερσαίο εκεί και βρίσκουμε ότι εκεί υπάρχει ιδιαίτερη ευπάθεια σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο, για το οργανωμένο έγκλημα εξετάζουμε μία σειρά παραγόντων Καταρχήν, αν ε, υπάρχει μια διαρκής απειλή από τη μια ομάδα, ζημία στην οικονομία, διαφθορά. Ε, των ε, επαγγελματιών όπως ε, παραδείγματο χάρη οι τραπεζίτες, σοβαρή ζημία, σοβαρή σωματική βλάβη και συνολικά υπάρχει μια περιγραφή εργασίας, δηλαδή να κερδίσουν χρήματα νομά και παράνομα και τα τελευταία 5-10 χρόνια είδαμε να αλλάζει το έγκλημα και ε, να μετακινείται περισσότερο από το οργανωμένο έγκλημα στη διεθνή σφαίρα. Για μας είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που να μην έχει και διεθνή διάσταση και αυτό μας ε, απέτησε να αλλάξουμε την τακτική μας και την απάντηση που δίνουμε. Πολλά έγιναν βάσει συνεργασία με άλλες διοκτικές αρχές και άλλες ομάδες που μπορούν να μας βοηθήσουν και συγκεκριμένα ε, έχουμε μια task force για το οργανωμένο έγκλημα, μια ομάδα κρούσης, ε, όπου ε, εκεί στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες διοκτικές στη Βορεια Ιρλανδία και επίσης συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στο Δουβλίνο και στην υπόλοιπη δημοκρατία της Ιρλανδίας να εξηγήσω τώρα τις ε, πληροφορίες ε, όπως τις κατανοούμε εμείς. Εδώ η κυρία πρόκληση είναι να ξέρουμε ε, όσα μπορούμε. Έχουμε τα συστήματα που μπορούν ε, να προσδιορίσουν τα γεγονότα, έχουμε τις διαδικασίες να αναλύσουμε και κατόπιν να ανταλλάξουμε, να λάβουμε δράση εγκαίρως. Και για να το κάνουμε αυτό μαζί με τις άλλες υπηρεσίες απαιτείται μια κοινή κατανόηση του προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Απαιτείται να οικοδομήσουμε μια πραγματική σχέση όπου να υπάρχει εμπιστοσύνη και να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγή πληροφοριών. εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό δεδομένη τη φύση ε, των πληροφοριών που ανταλλάσσουμε. Οι είναι ένα αγαθό και εννοώ ότι είναι χρήσιμο μόνο αν το μοιραζόμαστε οι ε, πληροφορίες δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά θα πρέπει να οδηγούν σε κάποια μορφή ποινική δικαιοσύνης επιβολής ε, της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για ένα άλλο αγαθό, δηλαδή προσπαθείς να προσπαθείς, ε, να ε, προβλέψεις ε, και να αποτρέψεις μελλοντικές δράσεις, δηλαδή δράσεις προληπτικά και εκεί κάνεις το καλύτερο για να εκτιμήσεις τι θα γίνει στη συνέχεια. Συχνά κάποιος αναζητά ευαίσθητες πληροφορίες που του δίνουν την ευκαιρία να χτυπήσει, δηλαδή να υπάρχει μια σύλληψη Παραδείγματο χάρη είναι ένα σπάνιο αγαθό, δηλαδή είναι δύσκολο να αποκτηθεί, μπορεί να είναι ακριβό, μπορεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, και απειλή της ζωής, αλλά επίσης πρέπει να επικεντρώνεται η συλλογή πληροφοριών ε, σε κάποιους ε, κανόνες που έχουμε στη διαδικασία και θα πρέπει να εξυπηρετεί και ένα σκοπό, όπως είπα. Και ε, τότε καθίσταται πληροφορίες ιδιαίτερα πολύτιμες σε σχέση με το τι θέλουμε να κάνουμε με αυτές. Όμως το καλύτερο είναι ότι αξίζει να ανταλλάζεις πληροφορίες με το τέτοιο και πάντοτε υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον. Όλοι λοιπόν προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε από κοινού το οργανωμένο έγκλημα. Τώρα εδώ θα σας δείξω την συνεργασία με την PSNI. Καταρχήν να πω ότι Είμαστε, έχουμε ένα και μόνο σύστημα, ένα νέο σύστημα πληροφοριών, γιατί είμαστε μία και μόνη αστυνομική υπηρεσία. Έτσι λοιπόν μπορούν όλοι να δουν το συνολικό σύστημα. Έχουμε ε, αποφύγει ε, να παραγωνίζουμε τις πληροφορίες, γιατί δεν ε, υπάρχει ουσιαστικά διαχωρισμός μεταξύ των διάφορων ειδών ε, πληροφοριών. δηλαδή, μιλάμε για εθνική ασφάλεια, για τρομοκρατία, οι κακοί δεν αναγνωρίζουν τις δικές μας περιγραφές εργασίας, δεν αναγνωρίζουν τους δικούς μας ορισμούς και εμείς πρέπει να είμαστε κάπου όπου να μπορούμε να παρέμβουμε όποτε έχουμε πληροφορίες και πρέπει να εκμεταλλευόμαστε ε, τις αδυναμίες τους. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα νέο σύστημα, δεν υπάρχουν στεγανά και αναλύουμε συνολικά μία ομάδα παραβατών. Μια, εδώ έχουμε μία σύντομη μελέτη που λέγεται επιχείρηση SLEEK ε, και θα σας ε, παρουσιάσω το ιστορικό το 2006 είχαμε μια επιχείρηση σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για να εντοπίσουμε ε, ένα πρόβλημα εμπορίας ανθρώπων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο λάμβανε χώρα τότε στην Βόρεια Ιρλανδία δεν μπορούσαμε να βρούμε πληροφορίες και πολιτικά στοιχεία ε, για την εμπορία ανθρώπων. Όλα αυτά άλλαξαν δύο χρόνια αργότερα όταν ε, ξεκίνησε η επιχείρηση ΣΛΗ και ήταν μια προδραστική έρευνα στην εμπορία ανθρώπων ε, και για τους σκοπούς της πορνείας. Ε, ε, τα θύματα ε, τα προσέλκυαν μέσω κάποιων αγγελιών που έβαζαν σε κινέζικο τύπο που ζητούσαν νταντάδες και υπήρχαν παραδείγματο χάρη εικόνες μιας οικογένειας έδειχναν οικογένεια που ζητούσε μια κυρία να προσέχει τα παιδιά τους και επίσης παρουσιάζονταν δουλειά σε γραφείο έτσι λοιπόν πίστευαν πίστευαν ότι θα έρθουν οι κοπέλες αυτές στην Βόρεια Ιρλανδία και θα έχουν ε, τη δυνατότητα μιας δουλειάς και εκπαίδευσης, όμως ήταν πραγματική βιτρίνα. Ε, ε, όταν ξεκινήσαμε το έργο μας το 2006, είχε γίνει η εμπορία ανθρώπων πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασιλείο και μετά είδαμε και στον τοπικό τύπο τέτοιες αγγελίες για συνοδούς και μέσω αυτού και μέσω ερευνών και πληροφοριών που συλλέξαμε αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι και εμείς έχουμε πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε διάφορες ε, πηγές πληροφοριών που συναντάμε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Χρησιμοποιήσουμε τους ε, υπαλλήλους στα λιμάνια και στα αεροδρόμιο και στα αεροδρόμια και ε, προσπαθούν ε, να δουν ποιο μετακινήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, παρακολουθούμε συγκεκριμένε μετακινήσει ανθρώπων και χρησιμοποιούμε και κάμερες κλειστού κυκλώματο, βίντεο κλειστού κυκλώματο από την ασφάλεια του αεροδρομίου και αυτό μα δίνει μια ιδέα για το ποια μπορεί να είναι η μετακίνηση. Επίση, όπω βλέπετε εδώ στην κορφή, Έχουμε συνεργασία με τις αστυνομικές υπηρεσίες, το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη ΣΟΚΑ ε, και επίσης συνεργαζόμαστε και με Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους και επίσης με τους γείτονες μας στο Δουβλίνο και με τις κινέζικες διοκτικές αρχές. Έτσι, λοιπόν, ε, μπορούσαμε να δούμε πώς μετακινούνταν τα άτομα από την Κίνα στο Δουβλίνο με πτήσεις και κατόπιν σε, δια της χερσαίας οδού περνούσαν στη Βόρεια Ιρλανδία και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι συνεργαστήκαμε με τις αρχές του Δουβλίνου και άλλους εταίρους. Επίσης, ε, προσπαθήσαμε να έχουμε και χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μετακινήσεις χρημάτων, αλλά και κάποιες εκθέσεις για... χρησιμοποίησαμε και κάποιες εκθέσεις για ύποπτη δραστηριότητα. Και φυσικά είχαμε και δική μας παρακολούθηση. Εδώ βλέπετε δύο χάρτες οι οποίοι ε, δείχνουν το μέγεθος της Βόρειας σε σύγκριση με την Ευρώπη και σε σύγκριση με τον κόσμο και είχαν στοχεύσει κάποιοι τη Βορεια Ιρλανδία για το οργανωμένο έγκλημα και φυσικά έχουμε ένα χερσαίο σύνορο που χρησιμοποιείται από το οργανωμένο έγκλημα για το όφελός του και αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς να συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους άλλους εταίρους στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στο Δουβλίνο. Αυτό είναι ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά έχει μια διεθνή λύση που είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και να βρίσκουμε τις ερευνητικές ευκαιρίες με τις άλλες υπηρεσίες διοκτικών αρχών. Το αποτέλεσμα συνολικά ήταν ε, ότι ανακτήθηκαν 10 πιθανά θύματα εμπορία ανθρώπων και αυτή ήταν η πρώτη μα επιχείρηση. Και αυτό είναι μέσω των δικαστηρίων. Αυτή είναι μια δημόσια παρουσίαση μια επιχείρηση που πέρασε και από τα δικαστήρια από τότε ανακτήσαμε άλλα 77 άτομα από την εμπορία ανθρώπων και έχουμε αναπτύξει κάποιες ε, ειδικέ ε, μεθόδους ε, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Βορεια Ιρλανδία και το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Χρησιμοποίησα αυτό ως παράδειγμα, γιατί υπάρχουν ε, κάποιες ε, πρακτικές ιδέες και αποτελέσματα που προκύπτουν. Το πρώτο είναι ότι το να είναι κάποιος ε, υπεύθυνο για την κλιματολογική ερευνά σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε στους υπαλλήλους μας κάποιες εναλλακτικές αξιοπλογές πρέπει να τους δίνουμε πληροφορίες για να μπορέσουν να δράσουν και το, για να το κάνουμε αυτό επιτυχώς κάποιος πρέπει να βλέπει τι συμβαίνει εντό αλλά και εκτός ε, της οργάνωσής του. Πρέπει να βρει με ποιου πιθανού εταίρους μπορεί να συνεργαστεί σε κάθε έρευνα και κατόπιν να αναπτύξει μια κοινή κατανόηση των απειλών να αναπτύξει μια ερευνητική διαδικασία μαζί τους, να συνεργαστεί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και να βρει ερευνητικές ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτεί. Αλλά ένα από το πιο σημαντικό είναι τα χρήματα. Πάντα πρέπει να παρακολουθούμε ακόμη και το τελευταίο λεπτό ε, του ευρώ γιατί ε, είναι ένας ε, τρόπος να δούμε τι γίνεται με την διοκτησία, και πρέπει να είμαστε προδραστικοί στο να οικοδομούμε σχέσεις. Επίσης, να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει δίσδυση στην οργάνωσή μας από το οργανωμένο έγκλημα και να μην έχουν διαφθαρή αστυνομική ε, που ασχολούνται με την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματο. Αλλά επίσης ε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το τι μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία. Έχουμε τους κατάλληλους πόρους, το κλειδί είναι η ανταλλαγή των πληροφοριών και να συνεργαζόμαστε για να συλλάβουμε τους κακούς. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Χάρης. Ε, το λόγο τώρα έχει ο κύριος ε, Όλιβερ το ο οποίος είναι επικεφαλής ε, των του κλιματολογικού στη Γερμανία και αυτός θα μας μιλήσει για το πώς χρησιμοποιεί η υπηρεσία του τις πληροφορίες ως ε, ένα σημαντικό στοιχείο. Εμείς το συζητήσαμε αυτό το θέμα και τις προηγούμενες ε, εβδομάδες και κάναμε για κάποιες διακρίσεις μεταξύ πληροφοριών, αποδείξεων και όλα όσα μπορούν να αφορούν μια αστυνομική έρευνα. 15 λεπτά έχετε κι εσείς για την παρέμβασή σας. Παρακαλώ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που, μου απευθύνατε. Ομιλώ εκ μέρους της Ενώσεως Γερμανών Εγκληματολογικών Υπαλλήλων που εκπροσωπεί τους ε, συναδέλφους μας από όλη την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Έχουμε 16 ομοσπονδίες, 16 αστυνομίες των ομόσπονδων κρατηδίων. Όλες μας διοχετεύουν αναλύσεις και αξιολογήσεις των δεδομένων. Επίσης έχουμε έρευνες από πανεπιστήμια, επίσης από ερευνητικά ιδρύματα αστυνομιών, που βέβαια όλοι αυτοί συμβάλλουν στην ίδια διαδικασία. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται ως εξής. Σκεπτόμαστε προς τα πίσω και σχεδιάζουμε προς τα εμπρός. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μια γενική αστυνομική γνώση για τις εγκληματικές δομές και δραστηριότητες και αυτό το θεωρούμε προϋπόθεση για την ε, δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Αναζητώντας έναν ορισμό της λεγόμενης intelligence στη Γερμανία, δηλαδή της συλλογής πληροφοριών, θα μπορούσα να σας πω το εξής. Η intelligence για μας είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα, ομάδες, δίκτυα, οργανώσεις, αλλά και γεωγραφικών εστιών εγκλήματος. Και εκεί παίζουν ρόλο και πολιτιστικά και πολιτικά γεγονότα. Βέβαια, η συνεργασία με την Αλοδαπή είναι ε, ένα από τα κυριότερα μέλημά μας. Στόχος μας είναι να αποκαλύψουμε παράλληλες κοινωνικές δομές στις οποίες ε, διαδικτυώνονται η, διαδικτυώνεται η εγκληματικότητα. Και επομένως και με προσωπικά δεδομένα, συλλογή και προσωπικών δεδομένων και άλλων που επιτρέπουν στην αστυνομία να διαπιστώνει τις τάσεις με τρόπο ρεαλιστικό και να ενημερώνει το πολιτικό επίπεδο. Μέσα στη διαδικασία αυτής της συλλογής πληροφοριών χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα Έχουμε για παράδειγμα την δομική ανάλυση η οποία εμβαθύνει στα προβλήματα και επιτρέπει να διατυπώνονται προτάσεις λύσεων για διάφορα προβλήματα. Την εναλλακτική δημιουργία ε, απεικονίσεων ε, και επίσης αναδρομική επισκόπηση. Χρησιμοποιούμε συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, τη μέθοδο Delphin δηλαδή, η οποία έχει και στρατηγική διάσταση. Για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία στο μέλλον. Επίσης, εξετάζουμε αποκλήσεις ε, επιπέδων και ούτω ε, Για παράδειγμα, για το διαδίκτυο, όπου είναι από αυτό το και μόνο το παράδειγμα προφανές ε, ποια είναι τα δεδομένα τα οποία ε, καλείται να αξιολογήσει η αστυνομία. Όπως είπε και σωστά ο κύριος Χάρης προηγουμένως, παρακολουθούμε και συνοδεύουμε και τις ανακριτικές και ερευνητικές διαδικασίες. Διεθνώς υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Εμείς έχουμε τις 11 φάσεις από τον καθορισμό του στόχου μέχρι την αξιολόγηση και οι αξιολογήσεις και αναλύσεις πρέπει να γίνονται με μια μεθοδολογία η οποία να μπορεί να είναι κοινή για όλους. Η ανάλυση βασίζεται σε πρότυπα αξιολόγησης για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα αλλά και να μπορεί να γίνεται και σε διεθνές επίπεδο. Για να λειτουργήσει η συλλογή πληροφοριών χρειάζεται ορισμένε προϋποθέσεις. Στη Γερμανία νομίζω έχουμε συμφωνήσει πάνω σε ένα ενιαίο επίπεδο προτύπων με σύγχρονη μεθοδολογία. Χρησιμοποιούμε κεντρικές υπηρεσίες όπου σειραίουν οι πληροφορίες και οι οποίες υπηρεσίες έχουν το καθήκον και είναι σε θέση να διοχετεύουν πληροφορίες και προς το εξωτερικό, αλλά και να δέχονται πληροφορίες τις οποίες να διοχετεύουν στο εσωτερικό. Άλλο σημαντικό είναι η στελέχωση. Χρειαζόμαστε αξιωματούχους οι οποίοι να διαθέτουν γλωσσικές ικανότητες, να έχουν κατανόηση των οικονομικών ε, εξελίξεων και του οικονομικού γίγνεσθε, γιατί είναι σημαντικό για να μπορέσει να μιλήσει, να μιλήσει κανείς πλέον για συλλογή πληροφοριών. Εκτός από αυτό χρειάζεται να θεσπίζονται ε, διεθνώς ισχυρά πρότυπα, να μιλούμε δηλαδή για τα ίδια πράγματα, να μιλούμε για τις ίδιες ε, πραγματικές περιγραφές εγκλημάτων, να αντιλαμβανόμαστε με κοινό τρόπο ποιος ενδέχεται να είναι ο υπεύθυνο μια εγκληματική δράση και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε επίσης πρότυπα για την αποθήκευση, χρήση και διαβίβαση ε, πληροφοριών και δεδομένων. Αυτά λοιπόν πρέπει όλα να γίνουν, να τυποποιηθούν, να γίνουν στάνταρτ. Είναι σημαντικό οι διαδικασίες αυτές να γίνονται σε βάση κοινών στάνταρτ, κοινών προτύπων, αυτά να μπορούν να ελέγχονται επίσης και ε, οι κεντρικές υπηρεσίες να είναι ενήμερε και για, και για το περιφερειακό γίγνεσθε και είναι επίση σημαντικό όταν οι, περι, ναι, οι περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες να γνωρίζουν ποια είναι τα αντικείμενα που απασχολούν άλλες ε, υπηρεσίες. Υπάρχουν λοιπόν εδώ σημεία τομής μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και κάποια αποτελέσματα συνέργειας. Καθώς επίσης και η διαχείριση των διαδικασιών στον τομέα ΟΚΑ. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να φτάσουμε, να, επιτύχουμε δηλαδή ένα επίπεδο ε, προτύπων που να είναι ικανοποιητικό. Γνωστό είναι επίσης ότι στα πλαίσια του λεγόμενου benchmarking γίνονται και συγκρίσεις διαφόρων υπηρεσιών για να δει κανείς που υπάρχει ακόμα δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξη αλλά και για να διδαχθούμε ημένα από του δε. Σημαντικό είναι, όπω είπαν και οι προηγούμενοι, στην διαδικασία συλλογή πληροφοριών να συμμετέχουν όλοι οι συνεργάτε Από τον αστυνομικό που κάνει την περιπολία, ο οποίο ενδεχομένω ε, συλέγει ε, προσωπικέ πληροφορίε ή τον αριθμό ενό αυτοκινήτου μέχρι την κεντρική υπηρεσία, η οποία ενο αυτοκινητου επεξεργαστεί την πληροφορία αυτή. Όλοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και γι' αυτό απαιτείται μια σοβαρή διαδικασία διαχείρισης των πληροφοριών, όπου όπως είπα να συμμετέχουν όλοι οι ε, συμμετέχοντες. Και εκεί βέβαια χρέος έχουν οι ε, κεντρικές υπηρεσίες να ενημερώνουν τους συνεργάτες τους. Το ίδιο ισχύει και για την περαιτέρω εκπαίδευση ή για διάφορες checklist που πρέπει να έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιούν ε, τους ε, υπαλλήλου μας, για παράδειγμα, για θέματα τρομοκρατίας και ούτω καθεξής. Το ίδιο σημαντικό είναι και η διαδικτύωση μεταξύ αστυνομία και ε, της οικονομίας. Police Private Partnership. Έτσι ώστε να εστιάζει η αστυνομία και σε προβλήματα τα οποία ακόμα δεν έχει εντοπίσει. Και να μην λησμονήσω και το δικαιικό πλαίσιο. Όπως είπε και ο κύριος Χάρης, εμείς ως αστυνομία στη Γερμανία είναι χωριστές ε, οι ε, λειτουργίες δίωξης. Πρέπει ωστόσο να έχουμε πάντοτε υπόψη μας όλες τις διαστάσεις, διότι χρειάζεται να συλλέξει η αστυνομία αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να σταθούν ενώπιον του δικαστού και βέβαια αυτά μέσα στα πλαίσια ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου. Μπορούν να ε, υπάρξουν και προβλήματα μέσα στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Είναι και ε, εγγενή αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, στην προκαταρκτική ε, έρευνα που λύγει η αρμοδιότητα της αστυνομίας, που αρχίζει η αρμοδιότητα των μυστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ε, παρακολούθηση πληροφοριοδοτών ή των λεγόμενων whistleblowers, αυτών που καταγγέλουν δηλαδή ε, πράγματα που υποπτύουν στην αντίληψή του στον χώρο εργασίας κλπ. Όλα αυτά χρειάζεται, χρειάζονται μια κοινή διαμόρφωση μέσα στα πλαίσια της κατανομής των καθηκόντων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ποια πράγματα μας απασχολούν εμάς ως επαγγελματική ομοσπονδία. Πρώτα-πρώτα η εικόνα της καταστάσεως που θα πρέπει να είναι αξιόπιστες. Επίσης, να καλύπτει και τις ε, ε, ζώνες, για παράδειγμα, στην, στο οικονομικό έγκλημα. Επίσης, η διαρκής παρακολούθηση, το follow-up, και μετά από την λήξη της ε, δικαστικής διαδικασίας ανάλυση της αποτελεσματικότητας της δράσεως των αστυνομικών αρχών. Και αυτό λοιπόν πρέπει να εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία. Εφόσον διαπιστώνονται αντικειμενικές αδυναμίες, είναι σημαντικό το intelligence process να φτάσει και στο επίπεδο της αστυνομίας, ώστε να εξαλειφθούν οι αδυναμίες. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησαν και οι προηγούμενοι. Η ΟΚΑ δεν σταματά. Το οργανωσμένο έγκλημα δηλαδή δεν σταματά στα σύνορα. Χρειάζεται επομένως συνεργασία των ε, αρχών και διεθνώς για τη συλλογή πληροφοριών και ούτω καθεξής. Και χρειαζόμαστε επίσης και στο ε, ευρωπαϊκό επίπεδο τη δημιουργία θεσμών και βέβαια η διαδικτύωση είναι το σημαντικότερο, διαδικτύωση δηλαδή των Ευρωπαϊκών Τραπεζών Δεδομένων πέρα από τα σύνορα. Για παράδειγμα, ε, πληροφορίες, δακτυλικά αποτυπώματα και ούτε καθεξής, που σίγουρα μπορούν να γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσει και να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας αλλά και να επεκταθεί περισσότερο για να αντιμετωπίσει ένα οργανωμένο έγκλημα που απλώνεται όλο και περισσότερο. Ε, σας ευχαριστούμε. Τώρα, η τελευταία εισηγήτρια ε, είναι η επικεφαλή τη ομάδα που είναι αρμόδια για την αστυνομική συνεργασία για τη σχέση με την Κυροπόλη και τη Κεβόλου, που θα μα μιλήσει για την ενδυνάμωση τη νομοθεσία και τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μα μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ανταλλαγή Πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σα μέρα. Είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή σας που μου δίνει την ευκαιρία σήμερα να έρθω και να ενημερώσω τους Ευρωβουλευτές για τα κύρια βρήματα του πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών για την επιβολή του νόμου που δημοσιεύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2012. Υπάρχουν δύο στοιχεία στο πακέτο αυτό. Το πρώτο είναι ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό μοντέλο συλλογής πληροφοριών που είναι γνωστό ως EXIM. Το δεύτερο στοιχείο είναι η έκθεση για την εφαρμογή της λεγόμενης απόφασης πριν. Μαζί τα δύο αυτά έγγραφα παρουσιάζουν την εικόνα της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών διασυνοριακά μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου, όπως επίσης δείχνει και ποιες είναι οι εξελίξεις και οι συστάσεις που πρέπει να γίνουν για τη συνέχεια. Εδώ θέλω να ξεκινήσω με κάποια ιστορικά στοιχεία. Το πρόγραμμα της Στοχόλμη ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις ανάγκες για να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό μοντέλο συλλογής πληροφοριών, ιδιαίτερα μετά από την αξιολόγηση της λεγόμενης Σουηδικής Πρωτοβουλίας και της απόφασης ΠΡΙΜ. Η ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Συλλογή Πληροφοριών βασίζεται σε μια προηγούμενη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2010, που παρουσιάζει μια εικόνα όσον αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών στον τομέα τη ελευθερία, τη ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Βασίζεται επίση και στην στρατηγική διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εσωτερική ασφάλεια που συμφωνήθηκε το 2009. Η πρόσφατη ανακοίνωση πάντως για το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Συλλογής Πληροφοριών βασίζεται στην συλλογή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου συμμετέχουν ειδικοί από τα κράτη-μέλη, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασιζόμαστε βέβαια και σε συζητήσεις με άλλους φορείς Όπω επίση και με όλε τι αρχέ για την προστασία των δεδομένων. Ποια είναι τώρα τα συμπεράσματα από την ανακοίνωση αυτή. Πρώτον, ότι η συλλογή πληροφοριών και ανταλλαγή πληροφοριών λειτουργεί πολύ καλά σήμερα και δεν υπάρχει λόγος να εισάγουμε νέα νομική βάση και νέα όργανα. Από την άλλη, αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμόζεται πλήρως, να εφαρμόζονται πλήρως τα εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και θα έρθω αργότερα στην απόφαση πριν. Πέρα από τις ε, συστάσεις που πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως τα κράτη-μέλη για την χρησιμοποίηση δηλαδή των ε, εργαλείων που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, την ε, Σουηδική Πρωτοβουλία και την απόφαση πριν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο έχει να κάνει με τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να παίξει το κανάλι της Europol. Λαμβάνοντα υπόψη μα του γενικού στόχου μα για συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιούμε το κανάλι αυτό τη Europol και το εργαλείο που είναι η ανακοίνωση Σιένα ως κεντρικό στοιχείο, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό θα μας βοηθούσε να αποφύγουμε καταστάσεις αβεβαιότητας όσον αφορά την επιλογή του καναλιού, κάτι το οποίο έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Και έτσι θα είναι πιο εύκολη η ανάμειξη της Europol όταν εμπίπτει στα πλαίσια της αποστολής της αυτό. Πράγματι, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο κανονισμό για την Europol, η πρόταση αυτή δηλαδή, βασίζεται μεταξύ άλλων στην ενίσχυση του ρόλου της υπηρεσίας αυτής ως κεντρικός άξονας. Και είναι γνωστό ότι η Europol είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας που πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο και πιο συστηματικά σαν στοιχείο για την ανταλλαγή πληροφοριών. Πέρα από αυτό βέβαια υπάρχει και η έννοια ε, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αστυνομικών ε, Αρχείων. Το 2012 ε, μελέτη που έγινε με τη βοήθεια όλων των χωρών μελών οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτά ήταν ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο έχουμε στοιχεία για κάποιον ο οποίος έχει αναμειχθεί σε ένα έγκλημα αν έχουμε στοιχεία του σε άλλα κράτη-μέλη. Από αυτή τη μελέτη λοιπόν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν χρησιμοποιηθούν σωστά και πλήρως τα εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, τότε αυτό το επιτυχάνουμε. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε είτε το σύστημα πληροφορών της Europol, είτε την ανακοίνωση Siena και βέβαια σε λιγότερο βαθμό την απόφαση Prüm και το σύστημα SIS2 που περιμένουμε. Βάσει λοιπόν του μηνύματος του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Συλλογής Πληροφοριών και βασιζόμενη στη σχέση ωφέλους κόστους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι το να δημιουργήσουμε αυτό το νέο εργαλείο έπρις δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή. Μια άλλη σύσταση είναι μέσα στα κράτη-μέλη να δημιουργηθούν κάποια ενιαία σημεία επαφής, τα SPOCs. Εφόσον υπάρχουν ε, τέτοια ενιαία σημεία επαφής, θα μπορεί να γίνεται πιο αποτελεσματικά ο συντονισμό κάθε φορά που σε διεθνέ επίπεδο ζητούνται κάποιες πληροφορίες. Τα σημεία αυτά επαφής δεν θα πρέπει να τα θεωρούμε βέβαια απλώ κάποια ε, κουτιά αλληλογραφία, κάποια κεντρικά mailboxes. Θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα υπάρχοντα κανάλια και να είναι εξοικειωμένα με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να έχουν ε, ως υπαλλήλους και συνεργάτες ε, άτομα από όλες τις αρχές ε, αρμόδιες για την επιβολή του νόμου που έχουν καταρτιστεί όμως βάσει του μελλοντικού σχεδίου κατάρτισης για την επιβολή του νόμου. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε, όλα τα, σε όλες τις βάσεις δεδομένων, βάσει φυσικά συγκεκριμένων κανόνων πρόσβασης. Τώρα το δεύτερο σκέλος του πακέτου είναι η έκθεση PRIM. Έχουν υπάρξει όμως πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και αυτό είναι κάτι πολύ θλιβερό ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι η προθεσμία για την εφαρμογή ήταν ε, ο Αύγουστος του 2011. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχει βελτιωθεί κατά πολύ κατάσταση, αλλά παραμένουν κάποια κράτη-μέλη που βρίσκονται πιο πίσω και που θα έπρεπε να επιταχύνουν το βήμα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η πλήρης εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη είναι κάτι αναγκαίο πριν προβλέψουμε ε, αλλαγές ε, στο νόμο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε υπάρχουσα στήριξη το Helpdesk για την απόφαση πριν, τη Europol, αλλά και άλλες δυνατότητες που προσφέρονται βάσει ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το Δεκέμβριο του 2014, μετά την μεταβατική περίοδο βάσει του πρωτοκόλου 36 της ηθίκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να προχωρήσει σε προσφυγές επί παραβάση. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα τα στατιστικά δεδομένα, είναι κάτι κεντρική σημασία στα πλαίσια της απόφασης πριν. Στο μεταξύ, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να μας βοηθούν να αξιολογήσουμε την προστιθέμενη αξία του μέσου. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε με το στατιστικό μοντέλο που έχουμε σήμερα. Όσον αφορά τώρα την στήριξη για τη λειτουργία του συστήματος, πιστεύουμε ότι το Help Desk ε, Prim στη Europol είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στη διάθεσή μας για αυτό το σκοπό. Στο μέλλον όμως μπορεί να υπάρχει ρόλος για την υπηρεσία πληροφορικής που είναι γνωστή ως Ευρωπαϊκή Ένωση Λίζα. Βέβαια αυτό πρέπει να το ξαναδούμε αφού γίνει η πρώτη αξιολόγηση της νέας υπηρεσίας που θα είναι το 2015. Τώρα στρεφόμενοι προς το μέλλον. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε κάποιες γενικές αρχές που πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών πάνω απ' όλα πρόκειται για την προστασία ε, του ιδιωτικού βίου. Επίσης το θέμα ε, της, ε, του ωφέλους και του κόστους της κάθε δράσης μας. Αλλά βέβαια πρέπει να επικεντρωθούμε και στην προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω για να επικεντρωθούμε στις πραγματικές μας ανάγκες. Αυτό υπογραμμίζει βέβαια και υπογραμμίζεται και στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Συλλογής Πληροφοριών και την έκθεση ΠΡΟΜ. Προκειμένου πάντως να γίνεται καλύτερο έλεγχος, προτείνουμε στην ανακοίνωσή μας να γίνεται ετησίως μία συζήτηση στα επίπεδα του ΚΟΖΗ που να είναι αφοσιωμένη στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόμου. Θα μπορούσε αυτό να γίνει ήδη στα τέλη αυτής της χρονιάς για πρώτη φορά και θα ήταν καλό γιατί έτσι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ανταλλαγή Πληροφοριών. Εννοείται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόμου δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Είναι όμω ο κύριο ε, τρόπο που, που έχουν στη διάθεσή του οι αρχέ των κρατών μελών για συνεργασία. Όλα τα εργαλεία είναι πολύ σημαντικά για να ενισχυθεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει το έγκλημα και βέβαια και την πιο σημαντική του μορφή που είναι το οργανωμένο έγκλημα. Εν κατακλείδη. Θα ήμασταν ευγνώμονε αν μα δίνατε την ευκαιρία να έρθουμε ξανά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σα ενημερώσουμε για τι μελλοντικέ εξελίξει και τα επιτεύγματά μα στον τομέα αυτό. Σα ευχαριστώ. Ε, εγώ σα ευχαριστώ. Τώρα να ξεκινήσουμε αμέσω με τη συζήτηση, να δώσουμε καταρχήν το λόγο στου συντονιστέ. Κυρία Ματιέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Δεν μπόρεσα δυστυχώς ε, να ακούσω την παρέμβαση του κυρίου Φαρσή. Λυπάμαι. Σημείωσα κάποια αρκετά θετικά σημεία, κυρίως ε, στην παρέμβαση του κυρίου Χάρης που ήταν πολύ συγκεκριμένη σε σχέση με την επιχείρηση ΣΛΙΚ, με το πώς έγινε η ανταλλαγή πληροφοριών και για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με τις τρίτες χώρες, με την Κίνα. Όμως έχω κάποιες ερωτήσεις. Τι γίνονται όταν φτάσουν τα δεδομένα, κυρίως με τα δεδομένα που έρχονται από μια τρίτη χώρα. Τι συμβαίνει, πώς τα διαχειρίζεστε, καταστρέφονται κατόπιν τα δεδομένα, για πόσο αποθηκεύονται. Μας ε, αναφέρατε και τις ποινές φυλάξεις για κάποια άτομα, όχι για όλα. Οι Κινέζοι που έμειναν στην Κίνα και τελικά είχαν ε, εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση εμπορίας ανθρώπων καταδικάστηκαν στην Κίνα και αυτοί που καταδικάστηκαν είναι αυτοί που καταδικάστηκαν από τα βαρλανδικά δικαστήρια. Αυτό κατάλαβα εγώ, αλλά υπήρχαν και καταδίκες στην Κίνα. Θα ήθελα να μου πείτε τι έγινε. Και έχω και μια ερώτηση για την κυρία Μίτσι Εξαιρετική η παρέμβασή σας. Μας την κατάσταση σε σχέση με την Europol. Όλοι είμαστε πεπισμένοι για τις πρόοδους που σημείωσε η Ευρωπολ και για το ότι πρέπει η Ευρωπόλη να είναι ακόμη πιο παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπηρεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, και για τη συλλογή πληροφοριών και όλοι εμπιστευόμαστε τη Europol, αλλά καθόλου δεν μας μιλήσατε για τη ΣΕΠΟΛ. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μας πείτε τι γίνεται σήμερα με τη ΣΕΠΟΛ και τι γίνεται με την κατάρτιση των αστυνομικών. Γιατί γνωρίζετε ότι η Europol ε, έρχεται αφού έχει λάβει χώρα το έγκλημα στο ευρωπαϊκό έδαφος, όμως και η κατάρτιση των αστυνομικών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και συμμετέχει και στην πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος ε, και θα ήθελα να αναφερθείτε κάπως σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε κύριε Ματιέ. Ο κύριος Κύρκο. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ε, προσκεκλημένους ομιλητές. Μία ερώτηση. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει για το θέμα της κατάσχεσης πόρων σημαντικών εγκληματιών. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των ομιλητών σχετικά με το ποια εργαλεία θεωρούν ότι χρειάζονται οι υπηρεσίες δίωξης για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον εγκληματικό τρόπο ζωής και την συμπεριφορά πολλών εκ των προσώπων αυτών που θεωρούν ότι είναι υπεράνω του νόμου και ιδιαίτερα για να τους πλήξουν βαριά σε αυτό που του ενοχλεί περισσότερο, στα περιουσιακά του στοιχεία δηλαδή. Τι πιστεύουν οι ομιλητές μας, ε, τι απόψεις έχουν ή τι έχουν ήδη εφαρμόσει. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Φαγιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα. Αυτό είναι το γεγονός, ούτε εθνοτικές διαφορές και ε, ξέρετε ότι σήμερα μετά την πτώση του σιδηρούν το παραπετάσματος έχει εξαπλωθεί και προς την Ανατολή. Μιλάμε για εμπόριο όπλων ε, κτλ. Φυσικά θα πρέπει οι διοκτικές αρχές να είναι ένα βήμα μπροστά από τους εγκληματίες, αναφέρετε κάποιες εξέχουσες πρακτικές ε, και τονίσατε κάποιες αδυναμίες, κάποιες ελλείψεις. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις ε, και θα αποφασίσετε εσείς ποιος θα απαντήσει. Καταρχήν, Χρειαζόμαστε πάρα πολύ σύγχρονες ερευνητικές ε, τεχνικές. Αναφερθήκατε στην κατάρτιση και στον εξοπλισμό για την καταπολέμηση του πιο σοβαρού εγκλήματος. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάποια συγκεκριμένα μέτρα, η κοινή κατάρτιση που θα μπορούσε να αναλυφθεί. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ενερμονιστεί σε αυτό το πλαίσιο, τι θα είναι πιο χρήσιμο. Δεν ε, αναφερθήκατε ιδιαίτερα στη σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Κανείς ε, δεν ε, ανέφερε το κέντρο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνό χώρο, το οποίο είναι υποσύσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι τέτοιες ειδικέ ομάδες, ε, ομάδες ειδικών, θα μπορούσαν ε, να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του οργανωμένου στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Ε, αν δεν καταπολεμήσουμε το κυβερνοέγκλημα, δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το έγκλημα γενικά σήμερα. Επίσης, η συνάδελφος αναφέρθηκε στη Σεπόλ και καθώς προερχόμαι από την Σλοβενία, να πω και κάτι ακόμα. Αναφερθήκατε στα τρίτα κράτη. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι άμεσο γειτονά μα. Αυτέ οι χώρε σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρηση. Η αντιπροσωπεία μα επισκέφθηκε τη Σερβία όπου ήδη είναι αρκετά αποτελεσματικές υπηρεσίες, αλλά θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να μου πείτε τι γίνεται με τη συνεργασία Συχνά μιλάμε για διαφθορά, για οργανωμένο έγκλημα, νομοποίηση παράνομων εσόδων ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Και ξέρετε και ότι η Σερβία είναι εστιακό σημείο. Πώς αξιολογείται λοιπόν την κατάσταση στις χώρες αυτές και ε, υπάρχει κάποια πρόοδος και πώς αξιολογείται τη συνεργασία σας με τις αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Μάλιστα, ο κύριος Νιτοντάν. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους τους Ομιλητέ και όλε οι ομιλήτριε δηλαδή που διέθεσαν τον χρόνο του γιατί ξέρω ότι είναι πολύ άσχολοι άνθρωποι. Ήταν δύσκολο να καταλάβω τι εννοείται γιατί οι διατυπώσεις ήταν πολύ προσεκτικέ και συγκρατημένε. και βέβαια η ε, συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται από το διαδίκτυο και επομένω σίγουρα δεν μπορείτε να ανοίξετε τελείω τα χαρτιά σα, Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Πάντω σα ευχαριστώ που ήρθατε. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε στην πραγματικότητα και οι συνάδελφοί μου το ίδιο πράγμα λένε. Ποιε είναι οι βελτιώσει που θα θέλατε να δείτε, που θα σα βοηθήσουν στη δουλειά σα, που θα σα διευκολύνουν στο μέλλον. Η Επιτροπή μα εξετάζει αυτή τη συνολική εικόνα τη Ευρώπη. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε εμεί ω Ευρωπαίοι. Αν δεν μπορείτε να το πείτε δημοσίω, στείλτε το μα γραπτά και θα το βάλουμε στην εκθεσή μα. Βελτιώσει δηλαδή που μπορούμε να σα βοηθήσουμε να επιφέρετε. Και πιο ειδικά τώρα, ρωτώ τον κύριο Χάρη, που ανέπτυξε με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ε, όραμα για την επιχείρηση SLEEK. Ποια ήταν η συμμορία αυτή, ήταν άνθρωποι από τη Βόρεια Ιρλανδία ή ήταν Κινέζοι οι οποίοι διείσδησαν στη Βόρεια Ιρλανδία και επομένως κατά πάσα πιθανότητα και άλλες χώρες ή ε, όπου στέλνουν δηλαδή οι Κινέζοι ανθρώπους γιατί η ηταν κινεζοι οι οποιοι διεισδησαν στη βορεια ιρλανδια και επομενως κατα πασα πιθανοτητα και αλλες χώρε οπου στελνουν δηλαδη οι κινεζοι ανθρώπου γιατι η κινα ε, έχω την εντύπωση ότι λειτουργεί μεθοδικά και αυτοί, αυτά τα 7 to 7 victims ήταν Κινέζοι θύματα. Με ενδιαφέρει να το μάθω. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν δηλαδή πολύ χρήσιμο που μας δώσατε ένα πρακτικό παράδειγμα, ένα παράδειγμα από την πράξη. Τώρα, προς τον κύριο Χουτ, ο Σουηδός συναδελφός μου που αναγκάστηκε να αποχωρήσει με παρακάλεσε να σας ρωτήσω το θέμα της ακαιρεότητας. Τι κάνετε για την Ιταλία όπου είναι διαβόητο ότι η Ιταλική αστυνομία ενδέχεται να έχει υπονομευθεί από εγκληματικά στοιχεία. Τι κάνετε σχετικά με αυτό, αν μπορείτε δηλαδή ε, να του απαντήσετε. Για την κυρία Αμίτσι, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε. Μία από τις ερωτήσεις που θα απασχολήσουν το Κοινοβούλιο είναι η πρόταση της Κομισιόν για την ε, προστασία της προσωπικής σφαίρας, data privacy. Γιατί χρειάζεται προστασία βεβαίως ε, των προσωπικών δεδομένων. Θυμούμε όμως που μίλησα με έναν Βέλγο αστυνομικό πριν από τα Χριστούγεννα, ο οποίος ειδικεύεται στο διαδίκτυο και μου είπε ότι αντιμετωπίζει το μέγα πρόβλημα ότι αν το παρακάνει στις έρευνές του κατά, κατά συμμοριών στο διαδίκτυο, τότε αναγκάζεται κάπου να σταματήσει για να μην παραβιάσει την προσωπική σφαίρα των εγκληματιών. Δηλαδή εκεί έχουμε καταλήξει, προστατεύουμε του εγκληματίες. Η ανησυχία δική μου είναι η Ευρωπόλ ίσως μέσω της Κομισιόν θεωρεί ότι πράγματι ενημερώνει τους ευρωβουλευτές, αλλά στο κάτω-κάτω εμείς θα νομοθετήσουμε σχετικά με την ανάγκη της επιβολής του νόμου, η οποία ίσως χρειάζεται κάποτε ε, να οδηγήσει στην άρση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ε, ε, το καθήκον μας είναι να προστατεύουμε τους πολίτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δίνουμε το ok στις διοκτικές αρχές να έρουν την προστασία αυτή. Είστε βέβαιοι ότι ενημερώνεται το Ευρωκοινοβούλιο επαρκώς για τις δύο αυτές πλευρές του νομίσματος, γιατί όταν θα προχωρήσουμε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, ίσως χρειαστεί να πούμε κάποια στιγμή, α όχι, καλύτερα ας προστατεύσουμε τους πάντες και τα πάντα και α αφήσουμε στην άκρη την επιβολή του νόμου. Τώρα, με του συναδέλφους μου έχω μιλήσει και άλλε φορέ για το έγκλημα και αυτό το νέο οργανισμό. Αύριο στις 8 προβλέπεται πρόγευμα που θα προεδρεύσω εγώ και θα είναι και ο πρόεδρος του Cyber, της Cyber Agency. Αν θέλει λοιπόν κάποιος να έρθει να ε, συζητήσει μαζί μας, πολύ ευχαρίστως να έρθει. Συγγνώμη, Μπίλ, ένα λεπτό. Εγώ ίσω δεν κατάλαβα καλά. Εγώ θα ήθελα όμω να μου διευκρινίσει κάτι για να δω αν εγώ παρανόησα την έννοια της ερώτησης ε, του Χολσμίτ ε, για την ε, Ιταλική αστυνομία. Δηλαδή μίλησες για δίσδυση στην Ιταλική αστυνομία, δηλαδή ε, ότι αυτοί δυσδύουν σε συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος για να διερευνήσουν αυτά τα εγκλήματα. Μήπως μπορείς να εξηγήσεις λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι από ποια χώρα προέρχεστε, από ποια χώρα μέλος προέρχεστε. Διακόπτη προέδρο. Όχι Μπίλ, εγώ δεν θέλω να υπερασπίσω τη δική μου χώρα, αν είναι έτσι. Απλώς ε, θέλω να υπερασπίσω του εκατοντάδε αστυνομικού που έχουν δολοφονηθεί στη χώρα μου. Γιατί αντιτάχθηκαν στη μαφία. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινιστεί κάπω καλύτερα το πλαίσιο. Είναι δύσκολο για μένα να το πράξω αυτό γιατί είναι ερώτηση του κύριου Σμιτ και ο κύριο Σμιτ έχει φύγει το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πριν από λίγα χρόνια είχα ηγηθεί μια αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού στο Παλέρμο και ακούσαμε εκεί από έναν Ιταλό αστυνομικό «Ε, είστε ασφαλεί που έρχεστε και συνεργάζεστε μαζί μας, αλλά μην πάτε να συνεργαστείτε με την άλλη αστυνομική δύναμη και έδειξε προ τα εκεί απέναντι, γιατί αυτοί έχουν υπονομευθεί από τη μαφία. Εσείς είστε Ιταλίδα και θα γνωρίζετε πολύ καλύτερα ε, αν είναι αληθές ή όχι αυτό. Εγώ απλώς μετέφερα ε, την ερώτηση του κ. Σμίτα αλλά φαίνεται πως έπεσα στη σφυκοφωλιά. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές ε, που παρευρίσκονται εδώ σήμερα το πρωί και μας εφηρώνουν τον χρόνο τους να ρωτήσω την κυρία Μίτση το εξή. Μιλήσατε γιατί το λειτουργεί καλά, αρκετά καλά η ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά όταν λέτε λειτουργεί λογικά, λειτουργεί τα καλά, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Τι περισσότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να λειτουργήσει καλύτερα ή έτσι όπως αναμέναμε. Και μιλήσατε για τα box, ε, δηλαδή για τα νέα σημεία επαφής και για τα γραμματοκιβώτια, τον email, μήπως μπορείτε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο στο τι σημαίνουν όλα αυτά και μιλήσατε και για κάποια κράτη-μέλη που καθυστερούν και ότι πρέπει να προχωρήσουμε και ότι και αυτά πρέπει να προχωρήσουν και να είναι πιο προδραστικά. Μήπως μπορείτε και εδώ να μας δώσετε περαιτέρω στοιχεία γιατί και ο Μπιλ και άλλοι είπαν ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε κάποιες συστάσεις και αν δεν έχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες, αν δεν ξέρουμε πώς να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, δεν μπορούμε και να βοηθήσουμε. Και νομίζω ότι ο Μπίλ πολύ σωστά αναφέρθηκε στο θέμα της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας και ο κ. Ε, θα πρέπει να τα γνωρίζει αυτά γιατί ε, ξέρετε ποιος είχε τα περισσότερα δικαιώματα τελικά το αθώο θύμα ή ο δράστης και φαίνεται ότι το, τα θύματα, τα δικαιώματα των θυμάτων ε, πολλές φορές ε, δεν λαμβάνονται υπόψη. Δηλαδή τα ξεχνάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και βλέπω ότι κάποιοι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, ότι κάποια πράγματα δεν συνέβησαν έτσι όπως έγιναν. Όμως, ε, να ρωτήσω τον κύριο Χάρης, που μας έδωσε ε, κάποια πολύ καλά παραδείγματα για μια επιχείρηση συνεργασίας ε, με την Κίνα ε, και μας είπε ότι είχαν στοχεύσει μια μικρή κουκίδα στο χάρτη, όπως η Βόρεια Ιρλανδία. Εμείς αυτό που κάναμε τόσα χρόνια είναι να έχουμε μια αστυνομική δύναμη που δέχτηκε πάρα πολλές επιθέσεις, αλλά θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι να γίνω τμήμα αυτού. σε ένα μεγάλο βαθμό ε, χρησιμοποιείται η περιοχή αυτή ως η πίσω πόρτα από που μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και τι γίνεται με την εμπορία εκεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Πόσο καλή είναι η συνεργασία για σας όταν πρέπει να περάσετε τα δικά σας σύνορα. Δηλαδή, πώς συνεργάζεστε με τη Europol και τη Eurojust, ε, συναντάτε γραφειοκρατία. Αναφερθήκατε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνη, ότι πρέπει να οικοδομήσετε εμπιστοσύνη με άλλες ε, δυνάμεις. Φαντάζομαι στους περισσότερους τομείς ε, αυτό είναι το βασικό, αλλά τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα και πώς ε, θα διευκολύνουμε τη δική σας ζωή καθώς ε, εσείς ε, είστε ένας αστυνομικός που αγωνίζεται για να πετύχει αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νίκολσον. Παρακαλώ κύριε Γιατόβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσεις χθες καθώς συζητούσαμε την έκθεση Ιακολίνο, μιλήσαμε πολύ για το ρόλο των τραπεζών στην ανταλλαγή πληροφοριών και σε ποιο βαθμό συνεργάζονται οι τράπεζες στην Ευρώπη αλλά και με τον ε, κόσμο γενικότερα. Ερώτηση προς τον κύριο Χάρης που τόνισε πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθούν οι αρχές τις ροές μετρητών. Και η δεύτερη ερώτηση για την κυρία Μίτσι. Τι γίνεται όταν, όταν γίνεται μια μεταφορά εγκληματικών δραστηριοτήτων και χρημάτων από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίθετο, από την Ένωση δηλαδή σε τρίτες χώρες. Γιατί γνωρίζετε ότι ε, ορισμένοι εγκληματίες χρηματοδοτούν ε, πράγματα σε τρίτες χώρες. Σάντρικα. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτο. Πρώτη, πρώτο θέμα δηλαδή. ποιο ρόλο παίζουν οι πληροφοριοδότες και για θέματα τρομοκρατίας είναι γνωστό είναι γνωστό ότι οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις των αρχών κατέσα δυνατές χάρη σε πληροφοριοδότες. Κατά πόσο λοιπόν χρησιμοποιείται το μέσον αυτό και στο οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν θετικές και αρνητικές εμπειρίες ενδεχομένως προετών στην Ολλανδία είχε υπάρξει είχε υπάρξει μια υπόθεση ε, λαθρέας εισαγωγής κοκαίνης σε κουτιά χυμών που είχε οργανωθεί από έναν Ολλανδό αστυνομικό μάλιστα Αν μπορείτε λοιπόν να επεκταθείτε λίγο για τα θέματα αυτά. Και επίσης σχετικά με την αξιοπιστία των εταίρων σε μια χώρα. Δηλαδή, οι αστυνομικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν καθαρά χέρια, να μην είναι διεφθαρμένες. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, είτε βρίσκεστε στη Γερμανία είτε βρίσκεστε στην Ιρλανδία και σκέφτεστε τι να κάνω, να δώσω τις πληροφορίες που διαθέτω στους Δανούς ή στους Έλληνες ή ούτω καθεξής. Πόσο ε, θεωρείτε ότι ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος αυτές οι πληροφορίες ε, να καταλήξουν τελικά στους ίδιους τους εγκληματίες οι οποίοι ενδεχομένως έχουν διεισδύσει στι αστυνομικές αρχές ή πληρώνουν κάποιου αστυνομικού και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει και εδώ να συζητηθούν κάποια μέτρα. Ποια εντύπωση έχετε αυτό πέστε μας. Είναι, είναι συγκεκριμένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα το, στο οποίο πρέπει να εγγύψουμε ή κατά τη γνώμη σας δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό ισχύει και για τις παλιές χώρες βεβαίως, αλλά και για τις σχετικά νέες χωρισμένε. Δηλαδή, με μια, ε, κατά κάποια, κατά, από μια άλλη άποψη, το πρόβλημα τώρα με ε, αλλεπάλληλες διευρύνσεις έχει ενταθεί. Μάλιστα, ο κύριος Μπορσελίνου έχει ζητήσει το λόγο. Κυρία, Η κυρία Μπορσελίνου, με συγχωρείτε. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές. Ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένα και δεν μπόρεσα να ακούσω τις παρουσιάσεις. Ε, δεν ήθελα να πάρω το λόγο γιατί δεν μου φαινόταν σωστό, αλλά άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση και από την ε, συζήτηση ήθελα να αναφέρω μια ιδέα που μου ήρθε στο νου. Δεν ε, μιλώ ως Ιταλίδα ή ως Ικελία, αλλά ως Ευρωπαία πολίτης. Άκουσα τις παρατηρήσεις ε, του Σουηδού συναδέλφου και πραγματικά εξεπλάγει γιατί αν αληθεύει κάτι τέτοιο εγώ νομίζω ότι πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη προσοχή Δηλαδή, αν μια αστυνομική δύναμη μιλάει για μια άλλη αστυνομική δύναμη, λέει μην ε, προστρέξετε σε αυτού ε, γιατί είναι διεφθαρμένοι. Εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σοβαρό, που δεν μπορούμε απλώ ε, με ένα χαμόγελο να βάλουμε στο αρχείο αυτό το επεισόδιο, γιατί ε, έγινε αυτή η παρατηρήση για το Παλέρμο και η Σικελία και το Παλέρμο είναι τοποθεσίες όπου έχει πληρώσει ψηλό τίμημα η αστυνομία. Ε, έχει, έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές και έχουν γίνει ε, πολλές θυσίες. ξέρω ποια είναι τα παλιά αστεία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων στην Ιταλία, μεταξύ των καραμπινιέρων και των άλλων αστυνομικών δυνάμεων, αλλά ίσως ε, στο παρελθόν αυτό να είχε λυθεί, να λύθηκε, ε, καθώς ο Φαλκόν ε, ανάγκασε αυτές τις δύο δυνάμεις, αυτά τα δύο σώματα να συνεργαστούν και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Είχαμε περιπτώσεις διείσδυσης, αλλά αντιμετωπίστηκαν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αλλά και με πολύ μεγάλο πόνο. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να εμβαθύνουμε σε αυτό που έγινε ίσως ε, κατά τη διάρκεια κίνηση της αποστολής στο Παλέρμο και αν υπήρχε πράγματι αυτή η δήλωση, εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτό να το περάσουμε έτσι και να το βάλουμε στο αρχείο. Ευχαριστώ κύριε Μπορσελίνο. Ναι, και εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, ε, να πω ότι έγιναν κάποιες πολύ σοβαρές αναφορές εδώ. Έτσι λοιπόν θα φροντίσω και εγώ να ρωτήσω προσωπικά τον κύριο Σμιτ, να του ζητήσω να είναι πιο ξεκάθαρος, να μας πει σε ποιο πλαίσιο έγιναν ε, κάποιες ε, τέτοιες κατηγορίες. Να σας πω ότι και εγώ δεν πήρα το λόγο επειδή είμαι Ιταλίδα ή Σικελή για να υπερασπίσω. Να με ξέρετε ότι μπορεί να ασκώ κριτική απέναντι στους μηχανισμούς της χώρας μου. Όμως εδώ μιλάμε για κάτι παραπέρα, γιατί αν μιλάμε για ένα γεγονός, ε, ε, η Ιταλική αστυνομία σε διεθνές επίπεδο χαίρει εκτίμησης από τις άλλες αστυνομικές δυνάμεις. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Και θα μιλήσω με τον κύριο Σμιτ ε, για να καταλάβω σε ποιο πλαίσιο έλαβε χώρα αυτό το γεγονό για να ξεκαθαρίσουμε μάλιστα ένα λεπτό, να τελειώσω και θα σας δώσω το λόγο και να κατανοήσουμε καλύτερα το σύνολο ο κύριος το έχει το λόγο πρώτα. I have to say, I think this... Ευχαριστώ, αλλά δεν έχει νόημα. Ειλικρινά. Υπάρχουν ερωτήσεις. Αν θέλετε εσεί να υποστηρίξετε την Ιταλία ή αν κάποιο θέλει να υποστηρίξει την Ιταλία, εντάξει, και εγώ μπορώ να το κάνω. Διαφθορά έχουμε και στη Δανία. Εσεί τι κάνετε τώρα, εμποδίζετε του ανθρώπου να απαντήσουν με ειλικρίνεια. Είναι γελίο. Όχι κύριε Σόντεργαρντ, ένα λεπτό. Δηλαδή εγώ πώς εμποδίζω να δοθεί απάντηση. Το λόγο θα το έχουν οι ομιλητές. Ε, απλώς ε, νομίζω ότι είναι παράλογο να εκτοξεύεται μια τόσο σοβαρή κατηγορία για οποιαδήποτε αστυνομική δύναμη γιατί είτε θα γίνουν κάποιες ε, κατηγορίες ε, με αποδείξεις, αυτό ναι, αλλά τώρα να λέμε ότι η Ιταλική αστυνομία είναι μια αστυνομία διαφερμένη, με συγχωρείτε, όχι επειδή είμαι Ιταλίδα, αλλά νομίζω κύριε Σαντέρκαρτ, εσείς χάσατε κάποιες παρεμβάσεις όπως κοκριτική, κριτική ε, απέναντι στους Ιταλικούς μηχανισμούς, αλλά μια τόσο έντονη κατηγορία νομίζω ότι πρέπει να αιτιολογείται. Εδώ δεν θέλει κανείς να κλείσει το στόμα σε κανέναν. Μάλιστα μπορούν ε, οι συγητές να παρέμβουν αν γνωρίζουν ε, τέτοια γεγονότα. Να μας το πούν. Εδώ ποτέ κανείς δεν έχει κλείσει το στόμα σε κανέναν. Ούτε βέβαια είναι η πρόθεση αυτής της Επιτροπής. Όμως, επαναλαμβάνω, απέναντι σε μια τέτοια κατηγορία και αναφορά θα πρέπει να εμβαθύνουμε, γιατί ε, να ζητήσουμε και περαιτέρω εξηγήσει από την Ιταλική αστυνομία. Επομένως, θέλω να περισπιστώ την αλήθεια και την πραγματικότητα. Παρακαλώ, κύριε Νιτοντάν. Well, just briefly. Πολύ σύντομα. Ο κ. Σόντεργατ έχει δίκιο. Έχουμε πολύ σημαντικότερα θέματα να συζητήσουμε. Θα επαναλάβω αυτό που είπα. Εγώ ηγήθη μια αντιπροσωπή, επίσημη αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ε, στη Σικελία, στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, για να εξετάσουμε πού εξαφανίζονταν πόροι τη Ένωση. Και μα είπαν Ιταλοί αστυνομικοί στη Σικελία, στην επίσημη αντιπροσωπεία μα. Αυτό που σα είπα προηγουμένω. Είναι γεγονό. Αν θέλετε λοιπόν μπορείτε να εξετάσετε και τα πρακτικά της ε, αντιπροσωπεία τη ε, επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και αυτά είναι δημόσια και υπάρχουν. Okay, grazie, Μάλιστα, βεβαίω θα το πράξουμε. Αλλά να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Έγιναν ε, κάποιες αναφορές ε, σε επιχειρήσεις, στην επιχείρηση στην Βορειοελλανδία με την Κίνα. Εγώ θα ήθελα να καταλάβω πέρα από αυτές τις επιχειρήσεις ε, το ίδιο τη σύνδεση μεταξύ των διαφορών κλιματικών οργανώσεων, μεταξύ των διαφορών μορφών ε, μαφίας. Και ε, τι κάλυψη έχουν τα δίκτυα αυτά, δηλαδή αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις και σε ποιο βαθμό. Και αν μπορείτε να κάνετε ένα κατάλογο αυτών των ε, εγκληματικών οργανώσεων ε, που είναι πιο ριζωμένες στην επικρατεία σας, που είναι πιο ισχυρέ. και σε τι δραστηριότητες επικεντρώνονται. Θα δώσω τρία λεπτά στον καθένα σας για να απαντήσετε. Με τον κύριο Φαρσί. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με κάποια στοιχεία στις ερωτήσεις σας. Θα αρχίσω από το πιο ευαίσθητο θέμα που είναι η διαφθορά. Ε, ναι, υπάρχουν ε, Ιταλοί αστυνομικοί διεφθαρμένοι, ναι, υπάρχουν Βέλγια αστυνομικοί διεφθαρμένοι. Και σίγουρα υπάρχει διαφθορά στην αστυνομία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι γιατί υπάρχει αυτή η διαφθορά και τι οδηγεί σε αυτή τη διαφθορά και την ε, συντηρεί. Ένα θέμα είναι τα μέσα, τα οικονομικά μέσα που έχουν δηλαδή οι εγκληματικές οργανώσεις. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το ιστορικό πίσω από το οργανωμένο έγκλημα, γι' αυτό συχνά μιλάμε για την Ιταλία, αλλά μαφίες δεν υπάρχουν μόνο στην Ιταλία, υπάρχουν και στα Βαλκάνια και αλλού. Υπάρχει και η μαφία των ασιατικών χωρών. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Από τη στιγμή όπου μία εγκληματική οργάνωση, και εδώ αναφέρομαι στο Βέλγιο, έτσι, στο λιμάνι της Ανβέρσας, έχει τη δυνατότητα 15.000 ευρώ να τα δώσει σε ρευστό, σε έναν τελωνιακό ή σε έναν αστυνομικό και στην περίπτωση εδώ σε έναν ε, λιμενεργάτη. Έτσι ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί και να επιτρέψει να περάσει η κοκαΐνη ε, μέσα από ένα κοντέινερ, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά μπορεί να αγγίξει τους πάντες. Πάρα πολύ λίγοι αντιστέκονται. Φανταστείτε έναν λίμεν ενεργάτη τι κερδίζει και του λένε «Κοιτάξτε, 15.000 ευρώ». Και τι σας ζητάμε στο κάτω-κάτω, απλώς το κοντέινερ αυτό που έχετε αναλάβει εσείς να μεταφέρετε, βάλτε το ανάποδα μόνο και μην το βάλετε ε, με το σωστό τρόπο, αλλά ανάποδα, τίποτα άλλο. Να λοιπόν ποιες είναι οι δυνατότητες για τη διαφθορά. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι υπάρχει διαφθορά οργανωμένη στα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πρόοδο. Ε, φυσικά πάντα μπορεί να δυσδύσει κάποιος ε, και να υπάρξει διαφθορά, αλλά προσέχουμε πάρα πολύ πώς προσλαμβάνουμε τους αστυνομικούς και υπάρχει και ολόκληρη σειρά μελετών και ερευνών που γίνονται ε, εκ των προτέρων, πριν δηλαδή προσλάβουμε έναν αστυνομικό. Είναι ένα πρόβλημα πάντως που πρέπει να έχουν ε, κατά νου όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες και να μην υπερβάλλουμε. Και γιατί, γιατί αυτό επηρεάζει και την διεθνή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς συνεργάζονται οι αστυνομικές αυτές αρχές και τι αξιοπιστία υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει εναρμόνιση των νομοθεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάνουμε αυτό σιγά σιγά. Από τη στιγμή που τα όργανα τα οποία υπάρχουν ε, τα χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη. Πριν αναφερθήκαμε στη Europol. Υπάρχουν τα κανάλια λοιπόν και άρα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Και από τη στιγμή που οι δύο δι' αυτοί υπάρχουν μέσα σε μια συγκεκριμένη δομή και με ευρωπαϊκή νομοθεσία, από εκεί και πέρα έχουμε ένα σωρό εγγυήσει για αξιοπιστία. Εννοείται τώρα ότι ο Ιταλός ή ο Γερμανός αστυνομικός που έρχεται σε επαφή με έναν Σλοβανό, Σολοβαίνο ή έναν άλλον τέλος πάντων συνάδελφό του, ε, εγγύηση για αξιοπιστία δεν μπορούμε να έχουμε 1100. Γι' αυτό και μιλάμε και για τους συνδέσμους που μπορούν να ενισχύσουν την διεθνή συνεργασία κάθε φορά που υπάρχουν ανταλλαγές μεταξύ των χωρών μελών. Πριν αναφερθήκαμε και στο μεγάλο πρόβλημα που είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο. Ε, θα συνεχίσουμε το μοντέλο που σας παρουσίασα πριν για το Βέλγιο. Το βασικό είναι η συμμετοχή των ανθρώπων. Γιατί υπάρχει αίσθηση στις αστυνομικές αρχές του Βελγίου τουλάχιστον ότι η διεθνής συνεργασία είναι θέμα ειδικευμένου προσωπικού, ειδικευμένων αξιωματούχων της αστυνομίας. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί η ανταλλαγή πληροφοριών είναι κάτι καθημερινό. Η πληροφορία αναλύεται και καταγράφεται καθημερινά από τις αστυνομικές αρχές. Άρα εδώ πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και αυτή είναι η προσέγγιση στην οποία αναφέρθηκα πριν. Να ευαισθητοποιήσουμε τους ε, αστυνομικούς που δουλεύουν επί τόπου, να συνειδητοποιήσουν ότι το έγκλημα είναι διεθνές, ότι οι εγκληματικές οργανώσεις περνάνε τα σύνορα με μια φοβερή ταχύτητα, αστραπής. Το Βέλγιο, για παράδειγμα, σε μια ώρα είναι κανείς από τη μια άκρη του Βελγίου στην άλλη και έχει ήδη μπει και στην ε, γειτονική χώρα. Τώρα όσον αφορά την ε, χρησιμοποίηση των δεδομένων. Για να βελτιωθεί η τροφοδότηση οργάνων όπως είναι η Europol, πρέπει να φτάσουμε στο στόχο που έχουμε τουλάχιστον στο Βέλγιο, να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή η μεταβίβαση των πληροφοριών στα διάφορα διεθνή όργανα να γίνεται σε χρόνο ντετέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μεταβάζουν την πληροφορία, εντάξει, ίσως όχι online, αλλά εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε τα impact projects στην Europol που επιτρέπουν η πληροφορία να μεταβάζεται με δυναμικό τρόπο. Έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματική όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Κάτι άλλο τώρα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Και εδώ χρειάζεται εναρμόνιση. Πρέπει να γίνει σε διεθνές επίπεδο. Αναφερθήκαμε πριν στις δυσδύσεις. Ε, ναι, και στους πληροφοριδότες. Ναι, προφανώς και αυτή η τεχνική της αστυνομίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Το Βέλγιο είναι μια μικρή χώρα και γι' αυτό ξέρουμε περισσότερο από οποιοδήποτε ότι μόνοι μας δεν θα τα καταφέρουμε. Χρειάζεται συνεπώς εναρμόνιση σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών αστυνομικών αρχών. Δεν είναι στο κάτω-κάτω κάτι καινούριο και παλιότερα τότε που ασχολιόμουν με επιχειρήσεις, μια από τις, πρώτη, πρώτες που είχαμε κάνει ήταν για την έκσταση. Με... Δυσδύσαμε τέλο πάντων στα δίκτυα για να μπορέσουμε να λύσουμε ε, το θέμα αυτό και να πιάσουμε τα εγκληματικά δίκτυα της έκστασης. Σιγά σιγά όλοι πρέπει να έχουμε μια αντίστοιχη νομοθεσία. κάθε χώρα από μόνη της, στη γωνίτσα της, είναι απομονωμένη και πώς να αντιμετωπίσεις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες είναι παντού στον κόσμο λίγο πολύ. Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω εδώ είναι θέμα, το θέμα του computer crime, το κυβέρνο έγκλημα. Εδώ υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία είναι η νομοθεσία πρέπει να τηρούμε κάποιες ε, αρχές που έχουν να κάνουν με την προστασία του ιδιωτικού βίου, των προσωπικών δεδομένων. Εντάξει, γι' αυτό δεν μπορούμε να μπούμε και να κοιτάξουμε τα προσωπικά δεδομένα όλου του κόσμου. Είναι θέμα δημοκρατίας και προστασίας του ιδιωτικού βίου. Από την άλλη όμως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Στα πλαίσια ε, διείσδυσης και undercover ε, δράσεων υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει και το European Crime Center που μας ε, επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές από το διαδίκτυο που εξελίσσονται συνεχώς. Είναι αδύνατον μία ομάδα ε, για το έγκλημα στο διαδίκτυο από μόνη της να μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία, αν μη τι άλλο, όσον αφορά την τεχνολογία για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε για όλες τις τεχνικές. Το clouding, για παράδειγμα, είναι μια τεχνική η οποία θέτει ζητήματα όχι μόνο τεχνικού χαρακτήρα, αλλά και προστασίας δεδομένων. Πού είναι η πληροφορία. Δεν είναι ούτε στην Αγγλία, δεν είναι ούτε στο Βέλιο. Ε, πού είναι. Είναι στο cloud, στο σύννεφο, στο νέφος αυτό. Μερικές φορές δεν είναι ούτε στο Βέλιο, ούτε καν στην Ευρώπη. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Χάρης για να απαντήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να αποσαφηνίσω κάποια θέματα σε σχέση με την επιχείρηση SLEEK και συγκεκριμένα τη συνεργασία με την Κίνα. Είχαμε διευκόλυνση από τη δική μας ε, υπηρεσία που είναι ένα βρετανικό, ένας βρετανικός φορέας ε, και αυτοί ε, μας διευκολύνουν με τους υπαλλήλους, τους ξεμετούχους στο Πεκίνο αλλά συνεργάζονται και με τους νομικούς επιτετραμένους εκεί και θεωρήσαμε ότι είχαμε καλή συνεργασία με την Κίνα. Επίσης συνεργαστήκαμε και σε περιπτώσεις δολοφονίας εμπορίας ανθρώπων και λαθρεμπόριο τσιγάρων. Σε ό,τι αφορά τώρα την απόδοση ποινών, υπήρξε ένας Κινέζο, υπήρχαν και μάλλον κάποιοι Κινέζοι, αλλά υπήρξαν και οι άνθρωποι που είχαν στήσει τη βιτρίνα ε, στην ε, Ιρλανδία έτσι λοιπόν υπήρχε και ένα τοπικό στοιχείο σε αυτή την επιχείρηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα χρήματα, η δίμευση περιουσιακών στοιχείων είναι πάρα πολύ σημαντική και η ποινική καταδίκη αλλά και η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων. Έτσι λοιπόν εκεί όπου έχουμε πληροφορίες για ένα άτομο και ε, για τον τρόπο ζωής του τον εγκληματικό που δεν εξηγείται σύμφωνα με τα έσοδα που δηλώνει και πιστεύουμε ότι προέρχονται από εγκληματικό τρόπο ζωής αλλά στις περιπτώσεις αυτές πολύ συχνά βλέπουμε ότι κάποιοι ε, φαίνεται στην Ιρλανδία να έχουν ένα ταπεινό τρόπο ζωής, αλλά όποτε πάνε στο εξωτερικό αλλάζει εντελώς το τρόπο ζωής τους. Έτσι λοιπόν ε, τα χρήματα πηγαίνουν σε υπεράκτιους προορισμούς και στην Βόρεια Ιρλανδία βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν ειδικές σχέσεις ε, με τις διοκτικές αρχές στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, γιατί πολλές ε, φορές προσπαθούμε να κατάσχουμε και περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν σε εκείνες τις χώρες. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Ιταλικές διοκτικές αρχές και το παράταμε αυτό εδώ και κάποια χρόνια και έχουμε κατανόηση για τις τελικές διοικητικές αρχές γιατί καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται υπό τρομερή πίεση αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με οποιαδήποτε ιδιωτική αρχή και αναφέρουμε πάλι στο ότι είναι σπάνιο αγαθό οι πληροφορίε γιατί είναι ακριβέ, είναι επικίνδυνο να τι βρει κανεί, είναι δύσκολο, κινδυνεύουν ζωέ κάποιων ανθρώπων για καλέ πληροφορίε. Πρέπει λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το, αυτοί που συλλέγουν τις πληροφορίες πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή και το πώς ε, τις ανταλλάσσουν. Έτσι λοιπόν, αν εμείς λάβουμε κάποιες πληροφορίες από του Ιταλούς, ε, πρέπει υπεύθυνα να το αντιμετωπίσουμε. Κάθε αστυνομική αρχή θα πρέπει να έχει στρατηγικές κατά της διαφθοράς και ένα τμήμα αυτού είναι ο έλεγχος των πληροφοριών εντός της οργάνωσης. Οι ευαίσθητες πληροφορίες θα πρέπει να ελέγχονται πάρα πολύ αυστηρά ως προς την πρόσβαση έτσι ώστε να μην δημιουργείται κανένας πειρασμός στους αστυνομικούς εκτός της έρευνας ε, επειδή θα γνωρίζουν παραπάνω θα πρέπει. Ε, αλλά επίσης ε, αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει ε, όσοι συμμετέχουν σε μία έρευνα να προσέχουν ε, με ε, ποιους ανθρώπους ε, συνευρίσκονται, ποιος είναι ο τρόπος ζωής τους, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, μπορεί να υπάρξουν πιέσεις και μπορεί να χρειάζονται κάποια χρήματα σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής κάποιου, σε σχέση με κάποια άλλα σημεία που αναφέρθηκαν. Εμείς ε, θεωρούμε ότι οι πόροι, οι ανθρώπινοι πόροι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις πηγές ε, των πληροφοριών. Αλλά όταν μιλάμε για μυστικούς αστυνομικούς ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη νομική ευθύνη του φορέα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις δικές μας ομάδες οργανωμένο κλίματος, δεν θα τις αποκαλούσα μαφιόζικες ομάδες. Θα δίσταζα να τις αποκαλέσω μαφιόζικες ομάδες. Ε, υπάρχει εσωτερική συνοχή και πειθαρχία. Πρόκειται για δύσκολες ομάδες και ε, βλέπουμε να υπάρχει έγκλημα που συνδέεται με τη μαφία ή με κινέζικες εγκληματικές ομάδες. Όμως όλα αυτά τα άτομα διαπράττουν κάποια εγκλήματα και πρέπει εμείς να μιχνεύσουμε τι συμβαίνει και να αναλάβουμε δράση και κάτι νομίζω που μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε είναι η ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων διασυνοριακά. Είναι δύσκολη η ανταλλαγή πληροφοριών, όμως τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούμε να τα ανταλλάξουμε, αλλά φαίνεται να είναι δύσκολη η νομική διαδικασία. Εμείς τι προσπαθήσαμε να κάνουμε πάντοτε, να επιταχύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών έτσι ώστε να φτάσουμε πιο γρήγορα στη δικαστική διαδικασία. Τώρα η διαδικασία μπορεί να διερκέσει μήνες και νομίζω ότι αν μπορούσαμε να έχουμε ένα streamline εκεί και αν είχαμε κοινέ έρευνες μέσω της Eurojust, θα έχουμε κοινέ έρευνε μέσω της Eurojust και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και επίσης είναι θετική και η περιοχή της Europol. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από μία θέση μη συνεργασία, μη ανταλλαγή πληροφοριών, μη συνεννόηση. Νομίζω ότι είμαστε σε μία καλή θέση. Απλώ ε, συνεχώ ε, θέλουμε να ζητάμε τρόπου βελτίωση, ακόμα και οριακού. Και αναφέρθηκε κάποιο και στα Βαλκάνια. Εμείς ε, στέλνουμε εκατοντάδε αξιωματικούς ε, στα Βαλκάνια. Τους στείλαμε, τους στείλαμε πριν 12 χρόνια ως ε, συμμετέχοντες σε μια αποστολή. Έχουμε ισχυρή σχέση μαζί τους, τους υποστηρίζουμε, τους παρέχουμε πληροφορίες, κατάρτιση κατά τη διαφθορά, στρατικές κατά τη διαφθορά, έρευνα για την καταπολέμηση σοβαρού εγκλήματος. Θα ήθελα να τονίσω ότι στα πλαίσια της συνεργασίας με έναν άλλο οργανισμό κάποιος είναι πάντα πολύ προσεκτικός με ποιον συνεργάζεται γιατί πρέπει να δει αν συνεργάζεται με τον σωστό άνθρωπο. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, αλλά έχουμε ήδη καθυστερήσει. Παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Χουτ θα είμαι σύντομο. Πρώτα, οι ροές, οι οικονομικές ροέ. Τέθηκε η ερώτηση ποια μέσα θα ήταν χρήσιμα ώστε να τραβήξουμε το χαλί κάτω από τα πόδια των εγκληματιών. Στο γερμανικό δίκαιο υπάρχει δυνατότητα να ανακτηθούν περιουσιακά ωφέλη τα οποία έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη ε, δράση. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα όταν ο τρόπος ζωής του κατηγορουμένου δεν συναρμόζεται με το δηλωμένο εισόδημά του, αφαιρείται το υπερβάλλον. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, δηλαδή ο κατηγορούμενος υποχρεούται τότε να αποδείξει την νομιμότητα των εισοδημάτων του. Αυτό βέβαια είναι ένα βήμα το οποίο ε, υπόκειται σε διάφορους δικονομικούς περιορισμούς. Ωστόσο είναι ένας τρόπος που μπορεί κανείς να λάβει υπόψη, διότι οι οικονομικές ροές διακλαδώνονται και διαδικτυώνονται όλο και περισσότερο διεθνώς. Ρωτήσατε επίσης ποιες είναι οι ενδεχόμενες βελτιώσεις που μπορεί να επιφέρει η πολιτική, το πολιτικό επίπεδο δηλαδή για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε καλό δρόμο. Οι θεσμοί είναι καλά εξοπλισμένοι. Έχουμε επαφές με την Ευρωπόλη. Υπάρχουν δυνατότητες επαφής με άλλες χώρες. Ωστόσο, το πεδίο είναι τεράστιο σε πόσες χώρες, για παράδειγμα, υπάρχει τυποποίηση των διατάξεων για την συλλογή των τακτηρικών αποτυπωμάτων. Το ίδιο υλικού DNA. Πώς μπορεί να εξασφαλίσει η γερμανική διοκτική αρχή ότι το υλικό DNA το οποίο έχει συλλέξει είναι συγκρίσιμο με το υλικό DNA που έχει συλλεχθεί σε άλλη χώρα. Είναι απαραίτητο λοιπόν ακόμα και για καθημερινά πράγματα όπως διαρρήξεις. Και, εκεί ακόμα υπάρχουν διεθνείς διασυνδέσεις και εκεί πρέπει να δραστηριοποιηθούμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο. Σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει κανείς πάντοτε να έχει υπόψη ότι χρειαζόμαστε βεβαίως ρυθμίσεις ως διώκτες που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες και από την ελεύθερη οικονομία. Επομένως, και για την διαπίστωση διασυνδέσεων μεταξύ των προσωπικών δεδομένων και των περισσοκών στοιχείων των διοκομένων. Για παράδειγμα, στις διάφορες χώρες μέλη είναι πολύ διαφορετικό ο τρόπο με τον οποίο μπορώ να διαπιστώσω ποιος είναι ο κάτοχος ενός κινητού τηλεφώνου. Χρειάζεται να συμπληρώσω 7-8 διαφορετικά έντυπα τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται και με ορισμένες νομικές διατάξεις. Ενώ σε άλλες χώρες αρκεί να πάρω ένα τηλέφωνο, να πετύχω το σωστό υπάλληλο και μου δίνει την πληροφορία αμέσως. Για την καταπολέμηση λοιπόν του οργανωμένου εγκλήματος χρειάζεται και η δυνατότητα να ρυθμιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα προσφεύγουν οι ε, διοκτικές αρχές και στην ελεύθερη οικονομία. Συζητήθηκε επίσης εδώ και η διαφθορά. Είναι όντως διεθνές πρόβλημα. Το ανέπτυξαν και άλλοι προηγουμένως. Σημαντικός παράγοντας είναι εδώ η σωστή στελέχωση, η σωστή μισθολογική αντιμετώπιση των ε, αστυνομικών που δεν πρέπει η μισθή τους να είναι τόσο χαμηλή που να μην τους επιτρέπει να συμμετέχουν δραστήρια στην κοινωνική ζωή. Πρέπει να, εξετάζονται, να εξετάζεται επίσης ποιοι πόροι έχουν χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δίωξη, με ποιον τρόπο διοχετεύονται οι πληροφορίες, αν ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος οι πληροφορίες αυτές να ε, διοχετευτούν σε ακατάλληλα πρόσωπα και ούτω καθεξής. Επίσης τέθηκε το ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριοδοτών. Και εδώ πρέπει να εξεταστεί και πανευρωπαϊκά ποια είναι η προστασία των πηγών των πληροφοριών. Πόσο βέβαιος μπορώ να είμαι ότι ο πληροφοριδότης μου εφόσον χορηγήσει πληροφορίε, θα είναι ασφαλής και δεν θα διωχθεί, για παράδειγμα, από άλλες ένομες ε, τάξεις άλλων χώρων μελών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τώρα για τα συμπεράσματα, κυρία Μίτση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα αυτό πρώτος η κυρία Ματιέ. Ναι. Είναι αλήθεια ότι εγώ δεν αναφέρθηκα στην ΣΥΠΟΛ στη σύντομη παρουσίασή μου και αυτό επειδή η ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό μοντέλο ανταλλαγής πληροφοριών καλύπτει τα εργαλεία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και πώς ε, γίνεται αυτή από τις αρχές που έχουν αναλάβει την επιβολή του νόμου. Η ΣΕΠΟΛ δεν έχει το ρόλο συλλογής πληροφοριών, είναι όμως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προκειμένου η αστυνομία και οι αστυνομικοί να αποκτήσουν τα προσόντα και το know-how για να κάνουν αυτή τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η ΣΥΠΟΛ είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό και ακριβώς τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις βελτιώσεις της υπηρεσίας όσον αφορά την ε, διαχείρισή της, την αποτελεσματικότητά της και τις επιδόσεις της. Η κατάρτιση αποτελεί μια πολύ βασική προϋπόθεση για να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών και ένα στοιχείο της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση των αρχών που επιβάλλουν τον νόμο. Και αποτελεί αυτό και αντικείμενο της επόμενης ανακοίνωσής μας που θα κάνει πιο συστηματική και θα προσφέρει νέα μυθολογία όσον αφορά την ε, συνεργασία μεταξύ την ε, κατάρτιση μάλλον για τη συνεργασία των ε, διοκτικών αρχών μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι οι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου να έχουν στην ε, διάθεσή τους την γνώση που τους χρειάζεται. Όπως είπε κάποιος προηγουμένως, δεν είναι θέμα ειδικού αξιωματούχου, όχι, είναι ο καθένας στην αστυνομία να γνωρίζει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για να υπάρξει αυτή η συνεργασία μεταξύ των ε, αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σημερινού εγκλήματος, του διασυνοριακού ιδιαίτερα εγκλήματος. Χρειάζεται επίσης να υπάρχει γνώση και κατάρτιση όσον αφορά τις προτεραιότητες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσει να καθορίζει. Η κατάρτιση λοιπόν για μας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συνεργασία μεταξύ αρχών που επιβάλλουν τον νόμο στις διάφορες χώρες. Αναφέρθηκαν τα SPOX, έτσι, τα ενιαία σημεία επαφής. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συνηθίζει αυτό, να χρησιμοποιεί τα αρχικά. SPOX λοιπόν. Η ιδέα αυτή του, των ενιών σημείων επαφής είναι η εξής. Θέλει η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών ε, μελών να είναι πιο αποτελεσματική. Και πιστεύει ότι αυτό θα επιτευχθεί εφόσον συγκεντρώνονται σε μία υπηρεσία οι αιτήσει αλλά και οι απαντήσεις για κάθε αίτημα όσον αφορά ανταλλαγή πληροφοριών. Κάποιες χώρες μέλη έχουν μια τέτοια οργάνωση ώστε να συγκεντρώνουν σε μια ενιαία υπηρεσία, σε ένα ενιαίο γραφείο, τους αρμόδιους για την επιβολή του νόμου των διάφορων υπηρεσιών. Στόχος τους είναι να συγκεντρώνουν κεντρικά όλα τα αιτήματα που γίνονται για τέτοιου είδους ανταλλαγή πληροφοριών. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, συμβαίνει αυτό. Αναφερθήκατε επίσης στην ε, προστασία δεδομένων. Βέβαια, ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας είναι ακριβώς η εφαρμογή υψηλών προδιογραφών προστασίας των δεδομένων. Αυτό βέβαια πρέπει να έχει να κάνει και με την επιβολή του νόμου. Εννοείται όμως ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάθε φορά τις ιδιαιτερότητες του χώρου και να φροντίζουμε να υπάρχει μια ισορροπία, ώστε οι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπορούν να φέρουν σε πέρα τα καθήκοντά του, προστατεύοντα βέβαια συγχρόνω τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των υπόπτων. Πιστεύω κι εγώ, όπως είπατε, πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται και να έχετε τη δυνατότητα όχι μόνο να ενημερώνεστε από τους ειδικού με ακρόσεις σαν τη σημερινή, αλλά αναφερθήκατε και στη Europol πριν. Πιστεύω ότι μπορείτε να καλέσετε την Europol να έρθει εδώ. Ναι, ναι. Και να σας δώσει πληροφορίες και να σας ενημερώσει για την καθημερινή ζωή της Europol όσον αφορά τη δίωξη του εγκλήματος. Κάποιος ε, ρώτησε κάτι για την ε, μεταβίβαση πληροφοριών προς τρίτες χώρες. Στόχος της ανακοίνωσής μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια υπάρχουν ε, διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες για ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά υπάρχει και η Europol η οποία συνεργάζεται με πολλές τρίτες χώρες. Και αυτό γίνεται μέσω συμφωνιών επίσημων συνεργασίας κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Λοιπόν, η, η Europol μπορεί να έχει ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες προς όφελος εννοείται των χωρών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ζήτησε το λόγο κύριε Χολμάιερ, παρακαλώ. Έχω μια ακόμη ερώτηση. Πριν λίγο καιρό είχαμε μία συζήτηση με αστυνομικούς εκπροσώπους από Τσεχία, Πολωνία, Γερμανία και μας είπαν ότι υπήρχαν κάποιες κοινές ερευνητικές ομάδες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος έτσι ώστε να πετύχουν πραγματική διασυνοριακή αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια όταν ζητάτε πόρους για τη συνεργασία αυτή. Μου είχαν πει ότι ε, η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική. Και ακούω ότι δεν ε, είναι αρκετά ευέλικτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προβάλλονται δυσνόητες ρυθμίσεις και δεν υπάρχει χρηματοδότηση ισομερής ίση για ε, διάφορες υπηρεσίες και αξιωματούχους. Να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο, είναι γνωστό ότι στα σύνορα προς Τσεχία υπάρχει η τριμερή συνεργασία Γερμανίας, Τσεχίας, Πολωνίας για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του σημαντικού λαθρεμπορίου ναρκωτικών αλλά και παραγωγή ναρκωτικών ουσιών. Σημειώνονται σημαντικά προβλήματα εκεί στη συνεργασία με το Βιετνάμ. Με ποιο τρόπο σκέπτεται να υποστηρίξει η Κομισιόν τι χώρε, έτσι ώστε να πιστεί το Βιετνάμ ε, να ε, γίνει πιο συνεργάσιμο και να μην μείνει μόνη της η Τσεχία για να αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά που της προκαλεί το Βιετνάμ με την παραγωγή ναρκωτικών ουσιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που αναφέρετε και τα προβλήματα που συναντούν στην πράξη πολλά κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Είναι κάτι που εξετάζουμε και θα θέλαμε να βρούμε κάποιους πιο ευέλικτους μηχανισμούς ε, για τη χρηματοδότηση ε, αυτών των ομάδων ε, στο επόμενο δημοσιονομικό πρόγραμμα αλλά φυσικά εξετάζουμε το πρόβλημα και θα δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την εκταμείευση των πόρων για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στις κοινές ερευνητικές ομάδες. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη ερώτησή σας, Θέλω να σας πω ότι δυσκολεύομαι τώρα να απαντήσω επί τόπου. Μήπως θα μπορούσαμε να το ξανασυζητήσουμε διμερώς και να σας δώσω πληροφορίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι, βεβαίω είναι η καλύτερη λύση. Ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους μας που παρευρέθηκαν εδώ σήμερα το πρωί. Τώρα θα ήθελα να καλέσω τους επόμενους ομιλητές να έρθουν εδώ στο βήμα της Προεδρίας. Τα Μάρα Μακαρέμπο, τον Πίτερ Κώστερς ε, που συνοδεύεται και από τον κύριο Πίτερ Φερκάουσεν.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 Ε, λοιπόν, εδώ έχουμε τον ε, τίτλο Σύνδεσμο μεταξύ τρομοκρατία και διασυνοριακού οργανωμένου κλίματο. Ε, κυρία Μακαρένκο, είναι εταίρο στη West Sands Advisory, η LLP, και θα μα παρουσιάσει μία μελέτη μεταξύ, για τον δεσμού μεταξύ των τρομοκρατικών ομάδων και των οργανωμένων κλίματο στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πίτερ Κώστερ είναι αρμόδιο για ε, τη επιχειρήσεις της Europol κατά της τρομοκρατίας ε, και θα μας μιλήσει για την ανάλυση της Europol για τη συνδέσεις μεταξύ οργανωμένου κλίματος και τρομοκρατίας. Η συζήτηση θα ξεκινήσει με το να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές για 15 λεπτά και θα ξεκινήσει η Ταμάρα Μακαρέγκο. Παρακαλώ. Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας αναφέρω τα συμπεράσματα της μελέτης μας για την σχέση του οργανωμένου εγκλήματος και με την τρομοκρατία. Η έννοια του Crime Terror Nexus είναι κάτι που υπάρχει πάνω από μία δεκαετία. Έχουν γίνει διάφορες αξιολογήσεις, αλλά δυσκολευόμαστε βέβαια να καταλήξουμε σε συγκεκριμένε τάσει, οι οποίες υπάρχουν, δεν υπάρχουν, στη σύνδεση ανάμεσα στο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αυτές οι δυναμίε ε, βέβαια οδηγούν στα εξή αποτελέσματα. Πρώτον, η σχέση μεταξύ των δύο αυτών φαινομένων δεν είναι τόσο ουσιαστική και άρα δεν την δίνουμε αρκετή σημασία. Και το δεύτερο, υπάρχει κατακαιρματισμός βέβαια της ε, αντιεγκληματικής στρατηγικής ή της στρατηγικής ε, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στις χώρες ε, μέλη. Η διασύνδεση έχει παραβλεφθεί για πολύ καιρό. Επίσης, κατά τη γνώμη μας, το δεύτερο είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι η σχέση αυτή υπάρχει. Ε, προσωπικά από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ασχολούμαι με την σύνδεση αυτή ανάμεσα στο έγκλημα και την τρομοκρατία και βλέπουμε ότι αυτή η σχέση ευδοκιμεί σε χώρους όπου επικρατεί αστάθεια. Ε, είτε είναι το Αφγανιστάν, είτε η Κολομπία, είτε η Λιβερία, είτε το Πακιστάν, είτε η Σιέρα Λεόν, αλλά όχι μόνο αυτά δεν μας ε, κάνουν εντύπωση. Το ίδιο συμπέρασμα βγάζουμε και αν κοιτάξουμε την περιφέρεια της Ευρώπης, σε περιοχές όπου επικρατεί η αστάθεια, όπως είναι τα Βαλκάνια ή ο Κάφκασος. Επειδή επικρατεί γενικά σταθερότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπόθεση ότι, το, ότι υπάρχει η σύνδεση αυτή είναι κάτι το υπαρχει η συνδεση αυτη αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό και δεν βλέπουμε ότι συχνά υπάρχει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις εγκληματικέ ομάδες και την τρομοκρατία μέσα στην Ευρώπη. Σχέση ανάμεσα στο εγκλήμα και την τρομοκρατία είναι πράγματα που παρεβλέπουμε. Όμως, πίσω από αυτό το σκεπτικισμό πρέπει να σκεφτούμε ότι τα, οι αποδείξεις που έχουμε τον τελευταίο καιρό δείχνουν ότι τελικά ε, υπάρχει αυτή η σχέση. Διότι προσαρμόζονται και οι εγκληματικές οργανώσεις και η τρομοκρατία, ώστε να μην είναι τόσο ευάλωτες και να μην μπορεί να βγαίνει προς τα έξω η σχέση που έχουν μεταξύ τους. Έχουν γίνει πολλές ε, μελέτες, δύσκολο βέβαια είναι να αποδειχθεί αυτό ξεκάθαρα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ε, ενδείξεις από πάρα πολλά παραδείγματα που πάνε προς την κατεύθυνση αυτή τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά όσο και στην περιφέρεια της Ευρώπης. Η μελέτη λοιπόν που κάναμε δείχνει ότι η σύνδεση αυτή είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο σε τρία επίπεδα, επιχειρησιακό, ε, σύλληψης σχεδίου αλλά και εξέλιξη στη συνέχεια. Υπάρχουν ε, αποδείξεις για τη σχέση σε επίπεδο σύλληψης σχεδίου ανάμεσα σε εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκρατικές. Αν τη σύνδεση αυτή δεν τη μελετήσουμε μεθολογικά και πολύ συγκεκριμένα, μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο για να κάνει τελικά το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία ένα φαινόμενο. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, τις ιδιαιτερότητες της σύνδεσης αυτής, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τα τελευταία χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύνδεση αυτή είναι είτε μεταξύ ομάδων, είτε μεταξύ δραστηριοτήτων. Πρέπει να καταλάβουμε την λεπτή διαφορά μεταξύ των δύο για να καθορίσουμε συγκεκριμένα τη στρατηγική μας. Η ασφάλεια που μας απασχολεί μέσα στην Ευρώπη σήμερα διαρθρώνεται βάσει 7 στοιχείων. Το πρώτο που αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί από άλλους είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρη η διάκριση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο, ανάμεσα στην νόμιμη και την παράνομη δραστηριότητα μερικές φορές και γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί. Δεύτερον, οι περισσότερες χώρες βέβαια αντιμετωπίζουν τους Ισλαμιστές τρομοκράτες σαν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά τους. Και αυτό ενισχύεται ακριβώ επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές τέτοιες τρομοκρατικές ομάδες δρούν μέσα στην Ευρώπη. Και ναι, μεν αποτελούν βέβαια τέτοια απειλή, αλλά υπάρχουν και πολύ περισσότερε εκτό Ευρώπη. Έπειτα, από τα Βαλκάνια. Πολλέ οργανώσει οργανωμένου εγκλήματο δρούν στα Βαλκάνια και ε, δυσδύουν όμω στι παράνομες αγορές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη σύνδεση επίσης με την Ανατολική Ευρώπη πρέπει να δούμε, γιατί εκεί έχουμε πολύ έντονο το φαινόμενο της εμπορίας ε, ανθρώπων. Έπειτα, οι νέες ε, προδιαγραφέ όσον αφορά την μετανάστευση δημιουργούν επίση τέτοια σύνδεση ανάμεσα σε διάφορες κοινότητε και τις ε, χώρες τους, κοινότητες της διασποράς ας πούμε και τις χώρες τους. Στην Ελλάδα για παράδειγμα. Πέμπτον. Υπάρχουν ε, επίσης συνδέσεις Αφγανιστάν, ε, Πακιστάν για παράδειγμα που χρησιμοποιούν και ανθρώπους που βρίσκουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομάδες ε, λοιπόν που, έχουν, ε, που ζουν στο εξωτερικό αλλά έχουν ε, σχέση με τις χώρες τους οδηγούν σε τέτοιες εγκληματικέ δραστηριότητε. Έπειτα υπάρχουν και νέοι τρόποι ε, εκπαίδευση των στρατευμένων αυτών ατόμων, Βόρειο Μαλή, Σομαλία ή Εμένη. Το βλέπουμε λοιπόν και στη σχέση Αφγανιστάν-Πακιστάν αλλά και στο Βόρειο Μαλή αλλά και αλλού όπου γίνονται απαγωγές Ευρωπαίων για να πάρουν μετά εγκληματικές αυτές οργανώσεις ε, λίτρα για να ελευθερώσουν τους ομήρους αυτούς. Στην Ινάμενας, ε, στην Αλγερία που ήταν αναμειγμένος ο Μουκτάρ ε, Μπερνγκουτάρ το είδαμε επίσης. Έκτον, η τρομοκρατία είναι ένα περίπλοκο βέβαια φαινόμενο με πάρα πολλά επίπεδα πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί με τα όπλα, με την ε, κατάρτιση αυτών των ε, εγκληματιών τελικά. Η ρύθμιση βέβαια που γίνεται, οι νόμοι που περνάνε, οι πιο αυστηρές προδιαγραφές, οδηγούν τους εγκληματίες να βρουν νέους δρόμους όμως. Καλό είναι δηλαδή που ενισχύουμε ε, τους νόμους, αλλά οι εγκληματίες βρίσκουν άλλους δρόμους. Έβδομο, ε, επειδή υπάρχει εξέλιξη βέβαια όσον αφορά την ασφάλεια, βλέπουμε ότι σε χώρες και σε περιοχές στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διαπιστώνεται μια σχέση μεταξύ των ε, γενναιών, ότι δηλαδή βάζουν μέσα στο παιχνίδι νέους, πολύ νέους, οι οποίοι νιώθουν καλά όταν στρατεύονται στην Ισλαμιστική ιδεολογία. Η έρευνα που κάναμε δείχνει ότι η σχέση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί διάφορες τυπολογίες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά ε, τις Ισλαμιστικές ομάδες ή εθνικιστικές ομάδες ή τους μεμονωμένους, μεμονωμένες ομάδες ε, τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει πάντα σχέση μεταξύ τους. Μερικές φορές, άλλες πάλι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες υβριδικές μορφές. Που ε, μπορεί να έχουν κοινά κίνητρα, για παράδειγμα, ή κοινή δράση. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει συμμετοχή και σε εγκληματικές οργανώσεις. Υπάρχουν πέντε απειλές από την σχέση οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, ε, φαίνεται ότι πολλές φορές γίνονται γάμοι συμφέροντος μεταξύ των δύο πλευρών. Το 2012 διαπιστώθηκε ότι, για παράδειγμα, η Ήρα ε, νομιμοποιούσε παράνομο χρήμα που ερχόταν από την Τραγκέτα στην Βόρεια Ιρλανδία. Και υπήρχαν επίσης και Ισλαμιστές ε, Ιταλοί που ε, συμμετείχαν με διασυνδέσεις στα Βαλκάνια. Έπειτα η συμμαχία μεταξύ των δύο που υπάρχει στα Βαλκάνια και στην περιφέρεια της Ευρώπης δημιουργεί νέα κίνητρα για ναρκωτικά ή για λαθρεμπορία ατόμων. Οι μεγαλύτερες απειλές ε, σήμερα από τον Κάφκασο στην Ευρώπη προέρχονται από ομάδες που είναι γνωστές ε, ότι δρούν χωρίς όρια. Ε, όπως για παράδειγμα το 2011 που είχαμε ομάδες Τσετσένων και Τούρκων που έκαναν επιθέσεις στην Ισπανία. Με συγχωρείτε, αν μπορείτε να διαβάσετε λίγο πιο αργά, τον διερμηνείς. Οι um, militant Islamist οργανώσεις χρησιμοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε ολόκληρη την ε, Ευρώπη και τη στήριξή τους. Το AQIM, για παράδειγμα, συμμετέχει στο εμπόριο ηρωίνης ε, μεταξύ Δυτικής Αφρικής και Ευρώπης. Έπειτα η Ελλάδα που βρίσκεται ανάμεσα στην Τουρκία και τα Βαλκάνια έχει μεγάλη σημασία για το οργανωμένο έγκλημα και προσφέρει δυνατότητες για την συνεργασία αυτή εγκληματιών και τρομοκρατών. Υπάρχουν όμως και τέσσερα απειλές κλειδί που αναδύονται από την σχέση αυτή στην Ευρώπη. Οι τρομοκράτες Ισλαμιστές καταφέρνουν και δυσδύουν πιο άμεσα στην εγκληματικότητα και την χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτήσουν τους σκοπείς τους. Έπειτα, ε, Βόρεια Αφρική και Πακιστάν, οι τρομοκράτες τους, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνται όλο και περισσότερο με το οργανωμένο έγκλημα για να χρηματοδοτήσουν τις τρομοκρατικές τους δραστηριότητες και σαν στόχους έχουν πρώτα τους Ευρωπαίους πολίτες που του απαγάγουν για λίτρα και έπειτα χρησιμοποιούν την Ευρώπη για να περνά τα ναρκωτικά τους. Έπειτα υπάρχουν πολλέ μορφές στη σύνδεση αυτή που δεν, ε, που δεν είναι συγκεκριμένα βάσει των μοντέλων των γνωστών που έχουμε μέχρι τώρα και το βλέπουμε αυτό και στο Αφγανιστάν και στο Ράκ. Έπειτα το θέμα της αστάθειας στην ε, Ευρώπη μερικές φορές, ορισμένε χώρες, κάνει την κατάσταση πιο περίπλοκη. Όπως σε χώρες που μόλις έχουν περάσει από πόλεμο. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε βέβαια την σύνδεση αυτή. Βλέπουμε ότι αντίθετα η σύνδεση αυτή οργανώνεται πάρα πολύ προσεκτικά και έχει σαν αποτέλεσμα να βελτιώνει τις, επιδόσεις τους, τις επιδόσεις τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η μελέτη μας έχει δείξει, έχει καταλήξει μάλλον σε διάφορες συστάσεις για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει και να αντιμετωπίσει τις απειλές από την σύνδεση αυτή. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς υπάρχει αυτή η σύνδεση και πώς εξελίσσεται μέσα σε μια συγκεκριμένη χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιος σήμερα το πρωί αναφερόταν στην ανταλλαγή πληροφοριών. Και... Όμως αναπεριφέρεια υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες στην εξέλιξη της μεθόδου αυτής. Πολλοί μελετούν το φαινόμενο παρόλο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε καλά πώς εξελίσσεται η σύνδεση αυτή και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει μία ενιαία λύση, είναι θέμα ανάλυσης ε, και των εγκληματικών οργανώσεων και των τρομοκρατικών για να δούμε τελικά πώς ε, συνδέονται κάθε φορά μεταξύ τους. Θα έπρεπε να υπάρχει μία μεικτή task force στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχύσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Οποιαδήποτε δουλειά που έχει να κάνει με τη σύνδεση των δύο πρέπει να λάβει υπόψη τη και διάφορες πολιτικές επιτυχίες. Όμως θα έπρεπε να υπάρχει μια νέα προσέγγιση απέναντι σε τρίτες χώρες, αν μη τι άλλο, για την σύνδεση αυτή. Οι προκλήσεις είναι συνεχιζόμενες, τώρα μάλιστα που έχουμε και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των υπηρεσιών που δρούν στα σύνορα. Ιδιαίτερα προτεραιότητα πρέπει να δώσουμε σε συγκεκριμένε περιοχές που πιστεύουμε ότι έχουν πρόβλημα. Οι περισσότερε δράσει των χωρών μελών επικεντρώνονται στην χρηματοδότηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αλλά πρέπει να δούμε και άλλες παραμέτρους στις ερευνές μας και να εντοπίσουμε και άλλα πράγματα πέρα από το αυτονόητο που είναι εγκληματικότητα, προσφέρει χρήματα στους τρομοκράτες. Η τάση πάντως των προσπαθών που γίνονται σήμερα να επικεντρώνονται σε ισλαμιστικές ομάδες μόνο δεν φτάνει τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν για διαφορετικές αλλαγές στις κοινωνίες τους, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς διάφορες ε, εθνικιστικές ομάδες ή μεμονωμένες ε, τρομοκρατικές ομάδες ε, προχωρούν στη σύνδεση αυτή με το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση μέσα στα κράτη-μέλη και πόσο σε περιφέρειες ολόκληρες και να καταλήξουμε σε μια στρατηγική για να αντιμετωπιστεί η διασύνδεση αυτή και να συμμετέχουν οι αστυνομικές αρχές, στρατιωτικές, να γίνονται και διπλωματικές προσπάθειες. Περισσότερη συνεργασία επίσης από τον ιδιωτικό τομέα είναι κάτι ουσιαστικό. Παρόλο που υπάρχουν αδυναμίες βέβαια στην ανταλλαγή πληροφοριών, το να αγνοούμε τη σύνδεση που όντως υπάρχει ανάμεσα στο έγκλημα και την τρομοκρατία ε, δεν μας βοηθάει να οργανωθούμε και να ε, ετοιμάσουμε νέες ε, τεχνικές αντιμετώπισης τους. Σε επιχειρησιακό επίπεδο τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ομάδες τους και οι υπηρεσίες τους που αντιμετωπίζουν το έγκλημα για την τρομοκρατία πρέπει να συνεργάζονται καταρχήν στην ίδια τη χώρα και μετά να προχωρήσουμε βέβαια και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος ε, Κώστερς, ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος της Europol για τις επιχειρήσεις, τις αντιτρομοκρατικές ε, και θα μας μιλήσει για την ανάλυση που γίνεται από την Europol για τη σύνδεση μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένων κλίματος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στην ΟΚΤΑ, ε, την ε, απειλή, αξιολόγηση απειλής οργανωμένου εγκλήματος, ε, όπου ίσως αναφέρεται ένα σύνδεσμος μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος πιθανόν αναφερά. δεν υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρο σύνδεσμος και τώρα ίσως να επαναλάβω κάποιο που είπε η κυρία προηγουμένως, στην ΟΚΤΑ 2011 γίνεται λόγο ε, για ε, διέλευση ναρκωτικών, ε, διακίνηση ναρκωτικών από την Αλκάιτα και το Ισλαμικό Μαγκρέμπ μέσω της Δυτικής Αφρικής. Και πάλι εδώ μιλάμε για τη διευκόλυνση της ε, δρομολόγησης των προϊόντων μέσω της Δυτικής Αφρικής. Επίσης ε, βλέπουμε ε, ότι υπάρχει και συμμετοχή της Ομαλικής Διασποράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να υπάρχει πιθανότητα χρηματοδότησης της Al Shabaab. Επίσης αναφέρονται ε, και στην πλαστογραφία εγγράφων ε, κτλ. Λεχθέντος αυτού, η τρομοκρατία είναι η άσχατη μορφή οργανωμένου εγκλήματος, ε, περιλαμβάνει κάθε είδους εγκληματικότητας και πάντοτε έχει και πολιτική συνιστόσα ή έχει πολιτικές επιπτώσεις. Ε, ε, ο στόχος ε, της τρομοκρατίας είναι η διαφορά που έχει ως στόχο με βία μέσα να φέρει ιδεολογικές αλλαγές. Και δεν μιλάμε εδώ για αυτοπλουτισμό. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ε, δεν θα μιλήσω για μονομένους τρομοκράτες και για την πιθανή του σύνδεση με τον οργανωμένο έγκλημα. Δεν θα μιλήσω δηλαδή για την περίπτωση του Νορβηγού, ε, ούτε στις αυτά που βλέπουμε στη Γαλλία. Θα μιλήσω για τρομοκρατικές ε, οργανώσεις η τρομοκρατικό έγκλημα είναι ένας κόσμος από μόνος του και σήμερα θα επικεντρωθώ στο θέμα της διακίνησης ναρκωτικών από τρομοκρατικές ομάδες η διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατία είναι εντελώ διαφορετικά διεγκλήματο εκ πρώτη όψεω. Όμω, πολλέ φορέ ε, τα δύο συνεπάρχουν πολλέ φορέ, ε, όπω ε, το άλογο και άμαξα. Αρχικά, οι τρομοκράτε και οι ήταν εχθροί των εμπόρων ναρκωτικών, γιατί οι γκερίλα τιμωρούσαν όσου εμπλέκουν εμπλέκονταν ε, σε διακίνηση ναρκωτικών. Ε, Όμω ε, είδαμε πολλέ φορέ τι οργανώσει να προβαίνουν σε διακίνηση ναρκωτικών και αριστερή και δεξιά ιδεολογία, αλλά και από άλλου, από οργανώσει που είναι υπέρ τη απόσχεση. Ο στόχο είναι να συλλεχθούν χρήματα για τι επιχειρήσει και πυρομαχικά. Τα χρήματα έχουν πάρα πολλέ χρήσει ανάλογα με τη φύση τη εγκληματική οργάνωση τα χρήματα μπορούν να ε, εξαγοράσουν μια υποδομή υποστήριξης που μπορεί ε, να προσφέρουν ε, και ακόμη και βοήθεια στις οικογένειες όσων των βοβιστών που συμμετέχουν σε επιθέσεις αυτοκτονίας. Πολλέ φορές τα χρήματα συλλέγονται και με νόμιμα και με παράνομα νέσα. Ε, επίσης καλωσορίζουν οι τρομοκράτες δωρεέ, από συμπαθούντες και πολλές φορές μπορεί να δηλώνουν ότι τέτοιε δωρεέ θα χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστικού λόγους, αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινό μυστικό ότι ένα ποσοστό των δωρεών θα χρησιμοποιηθούν για περισσότερο άμεσου τρομοκρατικού στόχου. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα χρήματα κερδίζονται με παράνομα μέσα, όπως η απάτη και άλλα εγκλήματα, όπως ε, και οι εκούσιες εισφορέ. κάποιε τρομοκρατικέ ομάδες έχουν εκστρατεία συλλογή ε, δωρεών ε, και ουσιαστικά υπάρχουν δωρεέ ανάλογα με το εισόδημα του καθένα και επίσης ε, μπορεί να επιτρέπουν και τη διακίνηση ναρκωτικών από διάφορε άλλε ομάδε, παίρνοντα ένα ποσοστό χρημάτων. Και αυτό καταλήγουν ε, ε, στα ταμεία των τρομοκρατικών ομάδων. Επίσης, ε, ε, τώρα η διακίνηση, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών είναι μία από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες στον κόσμο και μάλιστα τέτοιε ομάδες είναι καλά οργανωμένες, έχουν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και έχουν τα μέσα και την επιρροή να υλοποιήσουν τη δική τους δραστηριότητα. Ναι, να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά ε, ορισμένων τρομοκρατικών ομάδων. Βλέπουμε γιατί μπορούν να επωφεληθούν ε, από το εμπόριο ναρκωτικών γενικά. Ε, οι τρομοκρατικές ομάδες δεν είναι άμεση ανταγωνιστές στην αγορά ναρκωτικών με κάποιες εξαιρέσεις. Ένα άλλο μπόνους ε, για τους εγκληματίες είναι ότι οι τρομοκράτες αφήνουν λίγο χώρο στην αστυνομία να βρει πληροφοριοδότες. Επίσης, οι τρομοκράτες είναι άτομα που εμπιστεύονται οι εγκληματίες, γιατί και πάλι οι τρομοκράτες βασίζονται σε ιδεολογικά κριτήρια για τη δράση τους. Και τώρα η διαφορά μεταξύ εγκληματικών συμμοριών και τρομοκρατικών ομάδων ε, είναι ότι ε, είναι ε, περισσότερο ε, πιθανό, μάλλον λιγότερο πιθανό να υπάρχει προδοσία ή κακομεταχείριση των εγκληματιών από τους τρομοκράτες. Μια άλλη διαφορά είναι ότι γενικά τα κέρδη θα καταλήξουν στα ταμεία των τρομοκρατικών ομάδων ενώ με τους εγκληματίες αυτά θα καταλήξουν στις τσέπες τους και η έσχατη σχέση μεταξύ τρομοκρατών και εμπορίων ναρκωτικών βρίσκεται στην Νότια Αμερική και αναφέρομαι στην Κολομβία. Θεωρείται ότι η ΦΑΡΚ ε, εξαρτάται αποκλειστικά από χρήματα που προέρχονται από την παραγωγή και εξαγωγή κοκαίνης. Και τώρα εκτιμάται ότι η ΦΑΡΚ ελέγχει περίπου το 1 τρίτο ε, των εδαφών ε, της Κολομβίας. Κάποτε η Κούβα υποστήριζε στους αντάρτες με όπλα και χρήματα, αλλά αυτό σταμάτησε εδώ και καιρό. Το 98 οι αντάρτες είχαν ε, μεγάλες εκτάσεις που, όπου μπορούσαν ε, να κερδίσουν ε, πολύ περισσότερα χρήματα καλλιεργώντας κοκαίνη παρά άλλες καλλιέργειες. Έτσι λοιπόν πέτρεπαν στους αγρότες να καλλιεργούν κοκαίνη και ταυτόχρονα έλεγαν ότι αγωνίζονται για να έχουν ε, υψηλότερες αμοιβέ οι φτωχοί γεωργοί και ε, χρησιμοποιούσαν ένα μέρος του εισοδήματο ε, για την τρομοκρατία. Φυσικά μια άλλη περιοχή που μας ενδιαφέρει είναι η Μεσανατολή και η Κεντρική Ασία. Υπάρχουν ε, ε κάποιες αποδείξεις οι Σουνίτες Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ε, και ε, ακραίες ε, και ομάδες στο Λίβανο έχουν ενώ απαγορεύουν την ε, κατανάλωση οποίου ε, δεν απαγορεύουν την καλλιέργεια οποίου. Ε, Κάποιε τρομοκρατικέ ομάδες έχουν καταγγείλει ανοιχτά την χρήση ναρκωτικών ή έχουν συστήσει και πρόγραμμα κατά των ναρκωτικών. Παραδείγματο χάρη υπήρξε ε, στην Βόρεια Ιρλανδία το DAD, Direct Action Against Drugs, που θεωρείται ότι σχετιζόταν με το προσωρινό Ήρα και υπήρχαν ε, ε, μάλιστα και πυροβολισμοί, προσπαθούσαν να δολοφονήσουν κάποιους εμπόρους ναρκωτικών και ε, αυτή η ομάδα επίσης θεωρείται ότι ε, σε αυτήν την ομάδα υπήρξε δίσδυση ε, μέρους του προσωρινού Ήρα γιατί ουσιαστικά θεωρούσαν ότι αν έχουν μία στάση κάθε κατά των ναρκωτικών θα κερδίσουν τη συμπάθεια της κοινή γνώμης Προσπαθούσαν λοιπόν να ελέγχουν κάποιες περιοχές ε, και για όσο ο έμπορος ναρκωτικών υπάκουε τις εντολές ε, των τρομοκρατών μπορούσε να συνεχίσει την ε, δράση του. Είναι δύσκολο να βρούμε αποδείξεις για να αποδώσουμε εμπόριο ναρκωτικών στις τρομοκρατικές ομάδες. Πολλές φορές ένας εγκληματίας συλλαμβάνεται για Κάποιε ε, παραβάσεις σχετικά με τον νόμο ναρκωτικών και μπορεί να συνδέεται με κάποιες τρομοκρατικέ ομάδες, αλλά πώς να το γνωρίζουμε αυτό. Ε, σε κάποιε έρευνε, η πιθανή σχέση με την τρομοκρατία δεν έχει έλθει στο φως ή έχει παραμεληθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε τώρα με τη συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Διασδεμέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ τους ε, εισηγητές. Θέλω να αναφερθώ λίγο στο θέμα των σχέσεων ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Και θέλω πιο συγκεκριμένα να αναφερθώ σε ένα ιστορικό στοιχείο, ιδιαίτερο, που όμως διαρκεί. Είναι διάρκεια στο χρόνο. Και πρόκειται για το θέμα της ε, Κολομβίας που αναφέρθηκε έτσι αν πριν. Διαβάστε το βιβλίο του Ερμάν Κάστρο Καϊσέδο που παίρνει συνέντευξη από τον Παύλο Σκομπάρ και περιγράφει την προέλευση του λεφρεμπορίου ναρκωτικών και εξηγεί πώς τελικά δημιουργείται μια μεταμόρφωση, μια συγχώνευση αλλά και μια σύγχυση ανάμεσα στα ναρκωτικά και τη ΦΑΡΚ ή ανάμεσα στα ναρκωτικά και τον απελευθερωτικό στρατό. Με φοβερή βία ανάμεσα στα ναρκωτικά και το κράτος. Η ελαθρέμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν ε, φοβερά όπλα επίσης και τελικά ένας Ισπανός και Βάσκος γνωστός εισήγαγε την τεχνική των εκρηκτικών σαν ε, μέσο που χρησιμοποιούν ε, οι λαθρέμποροι ναρκωτικών. Ήμουνα στο Κάλι την προηγούμενη εβδομάδα στην κοιλάδα του Κάλκε που πάντα είναι καυτή περιοχή όσον αφορά τις θροπραξίες. Πολλές. Εκεί υπάρχουν οι ΦΑΡΚ, υπάρχουν οι λαθρέμποροι ναρκωτικών, η Βάκριμ και η παραστρατιωτική. Και δεν υπάρχει τρόπος να εντοπίσει κανείς ξεκάθαρα που χωρίζονται μένα από τους δε. Όμως υπάρχει συνεργασία, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Και είναι επίσης αδιαφυσβήτητο ότι υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Και αυτό μάλιστα και από ένα πρόσφατο γεγονός, πάρα πολύ σκληρό, που έλαβε χώρα στη δικιά μου, τη χώρα, στο δικό μου το κράτος, το Μάρτιο. Αυτά τα σχόλια είχα να κάνω για να συνεισφέρω και εγώ κάπως στη συζήτηση. Γιατί Η περίπτωση της Κολομβίας είναι χαρακτηριστική για αυτά που συζητάμε. Υπάρχουν φυσικά και άλλες ποικιλίε και άλλες περιπτώσεις στη Τσιχάτη αλλού με άλλες μορφές συνεργασίας στο Βόρειο Μαλί, βορείος του Τουμπουκτού δηλαδή. Είναι σαφές ότι υπάρχει. Αυτό το σχόλιο είχα να κάνω. Ευχαριστούμε κύριε Δίας Δεμέρα για τις ενδιαφέρουσες σκέψεις. Ο κύριος Νιτοντάν. Ευχαριστώ και τους δύο προσκεκλημένους πραγματικά σαν να παρακολουθούσα κινηματογραφική ταινία έντονης δράσης. Ελπίζω να μας δώσετε αντίγραφα των ε, παρεμβάσεων τους, γιατί ήταν τόσο περίπλοκα και πυκνά τα κείμενά τους που δεν μπόρεσα καν να παρακολουθήσω, κι ας ήταν αγγλικά και η μητρική μου γλώσσα είναι τα αγγλικά. Το ερώτημα είναι, τι να συστήσουμε εμείς η δική μας Επιτροπή για βελτίωση της κατάστασης. Αν θέλετε να πείτε κάτι τώρα ή να μας το διαβάσετε αργότερα θα μας βοηθήσει πολύ για τα συμπεράσματα της εργασίας της Επιτροπής μας. Πάντως έχω και ορισμένα επιμέρους ερωτήματα για τον κύριο Κώστερς. Κερδίζουμε ή χάνουμε στον αγώνα αυτό. Απλή ερώτηση. Κερδίζουμε απέναντι στους κακούς ή κερδίζουν αυτοί για την κυρία Μακαρένκο. Κοίταξα λίγο στο Google να βρω την εταιρεία σας που δεν την έχω ξανακούσει ποτέ και χρησιμοποιώ και Safari και Google και η ιστοσελίδα σας αδύνατον. Δεν ανταποκρίνεται, δεν ανοίγει. Βλέπω άλλα για το West Sands, αλλά η δική σας είναι απόλυτα κρυμμένη. Έχετε ιδέα, το γνωρίζετε αυτό. Και δεύτερη ερώτηση. Τι πάει να πει nexus. Χρησιμοποίησατε πολύ συχνά τη λέξη νέξους που σημαίνει σύνδεσμος ή κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται να είναι κάποια ειδική ορολογία. Τι πάει να πει νέξους. Ε, Για εξηγήστε μας, είναι πολύ σημαντικές προχωρήσεις που μας δώσατε, αλλά τουλάχιστον τις καταλάβουμε. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να δώσω το λόγο στους εισηγητές. Παρακαλώ, κύριε Μακαρένκο. Ευχαριστώ. Πολλές οι ερωτήσεις. Για τα σχόλια για την Κολομβία, μάλιστα, τα λάβαμε και φυσικά πολλές φορές ε, η Κολομβία ε, χρησιμοποιείται ως περίπτωση μελέτες για να δούμε πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Ε, δίνει ένα καλό παράδειγμα και μας βοηθά να μάθουμε όμως ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει εδώ και δεκαετίε αυτή η σχέση στην Κολομβία μεταξύ τρομοκρατία και εμπορών ναρκωτικών και εγκληματιών. βέβαια, παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι έχουμε ε, μεταφέρει τις εμπειρίες αυτές σε άλλα μέρη του κόσμου. Σας ευχαριστώ που το αναφέρατε λοιπόν και το σήμασα με Τώρα, οι ερωτήσεις για το τι κάνει η Επιτροπή ποιες θα ήταν οι συστάσεις που θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή για να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα σας παραπέμψω σε αυτή τη μελέτη που εκπονήσαμε, γιατί πρόκειται για ένα σύνολο συστάσεων και δίνει και κάποιες ε, διευκρινήσει σε σχέση με τα συμπεράσματα που σας παρουσίασα σήμερα με μεγάλη ταχύτητα και ζητώ συγγνώμη που μίλησα τόσο γρήγορα. νομίζω ότι μιλούσα αργά αλλά τέλος πάντων ζητώ συγγνώμη. Έχουμε διάφορες συστάσεις σε αυτό το έγγραφο και ελπίζω ότι θα σας βοηθήσουν. Τώρα, αν θέλετε περαιτέρω διευκρινήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Τι σημαίνει η ώρας νέξου, σύνδεσμος. Και πάλι ορίζεται στο έγγραφο ο Nexus είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Εγώ δημοσίευσα αρχικά ένα άρθρο μεταξύ της, για τη σχέση οργανωμένου εγκλήματος ε, και τρομοκρατίας το 1998 και σε αυτό το σύντομο άρθρο, μετά από χρόνια έρευνας επιτόπου, εφόσον με ενδιαφέρε το ζήτημα, κατέληξε σε ένα αρχικό μοντέλο για το πώς η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα αλληλοσχετίζονται. Και στα σχόλιά μου Αναφερθήκα σε έναν ε, οργανωτικό, σε έναν επιχειριακό, επιχειριακό συνδυσμό και σε έναν εξελικτικό συνδυσμό. Ο οργανωτικός συνδυσμός είναι αυτό, μία σχέση μεταξύ δύο ξεχωριστών οργανώσεων. Έχουμε μία, οργάνωση, ε, μία ομάδα οργανωμένου εγκλήματο και μία τρομοκρατική ομάδα. Δηλαδή ένα πυρήνα ισλομιστών, παίρνουμε το εδώ και την τραγκέτα και οι δύο ξεκινούν μια συναλλαγή. Ε, τώρα, δεύτερο επίπεδο σύνδεσης ε, είναι αυτό που αποκαλούσαμε επιχειρησιακό, δηλαδή οθετήση των τακτικών του άλλου. Και ο κύριος Διαδεμέρα ανέφερε την Κολομβία και οι ίδιοι έμποροι ναρκωτικών ε, να χρησιμοποιούν οι ίδιοι βόμβες για να έχουν πολιτικό αντίκτυπο στο τότε οι ε, αρχές ε, άρχισαν να δυσδύουν ε, σε αυτούς. Έτσι λοιπόν έχουμε τις τακτικές που χρησιμοποιούν ε, οι τρομοκρατικές ομάδες και έχουμε από την άλλη τους τρομοκράτες που να υιοθετούν εγκληματικές πρακτικές. Και όταν ε, μιλάμε για την ε, χρηματοδότηση τρομοκρατία, τρομοκρατίας, αυτό είναι μαλά, δείτε πιο συγκεκριμένε εγκληματικέ ε, δραστηριότητες. Έχετε τους Τίγρη Ταμίλ, που έχουν προβεί και σε εγκληματικές πρακτικές όπως εκβιασμούς, απαγωγές και έχουν τέτοια δίκτυα. Και τέλος έχουμε το σύνδεσμο τον εξελικτικό. Αυτός είναι κάπως πιο πολύπλοκος και εδώ είναι φιλός μας ο χρόνος. Αρχίζουμε να εξετάζουμε ομάδες όπως η ΦΑΡΚ που έχουν ξεκάθαρη πολιτική στρατηγική, βασίζονται στην ιδεολογία. Αν δείτε την αλλαγή ε, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, μπορείτε να δείτε σήμερα ότι οι ΦΑΡΚ είναι πιο εγκληματικέ στη φύση τους παρά τρομοκρατικές. Βέβαια μπορούμε να μιλάμε αιωνίω γι' αυτό και εγώ θα επιμένω και εγώ προσπαθώ να βοηθήσω την Κολομβία να κατανοήσει το ΦΑΡΚ γιατί πρόκειται για εγκληματική οργάνωση και καλλιεργούν παπαρούνες στα σύνορα με το Περού. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ε, για μένα αυτό ότι δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία. Έτσι λοιπόν ε, βλέπετε ε, την εξέλιξη, αν δείτε και τι συμβαίνει με το ΠΚΚ και το KLA. Και Βλέπετε, πολλές φορές υπάρχει εξέλιξη, μερικές φορές αλλάζει επιχειρησιακή στρατηγική, αλλάζει ηγεσία, μπορεί να στρατολογήσουν κάποιους ανθρώπους που δεν γίνεται βάση ιδεολογίας ε, η στρατολόγηση αυτή, αλλά τους πληρώνουν. Έτσι λοιπόν, ε, γι' αυτό χρησιμοποίησα τον όρο Nexus, γιατί περιλαμβάνει πολλά στοιχεία. Uh, Για την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μου μέχρι το βράδυ ήταν ε, διαθέσιμη, τώρα έχει πέσει. Ε, γιατί ε, την εξυγχρονίζουμε τη σελίδα, έτσι λοιπόν μάλλον είναι κακή στιγμή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστερς. μπορεί να απαντήσει και μπορούμε να δώσουμε και το λόγο και στο συναδελφό του. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση ήταν ποιες συστάσεις κάνουμε προς την κατεύθυνση της Επιτροπής σας ή ποιες να κάνει να χρησιμοποιήσουν σωστά τα εφιστάμενα μέσα και τους εφιστάμενους διάβλους επικοινωνίας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με όλο το σεβασμό που σας έχουμε, έχουμε εργαλεία. Μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα, πάντοτε βέβαια, αλλά αυτά που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας θα πρέπει να αρκούν κανονικά για την αντιμετώπιση των καθημερινών καθηκόντων μας. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ευρωπόλ αναζητούμε συνεργασίες με την κοινότητα της intelligence Άρα, συστάσεις θα κάναμε εμείς για πιο στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών και των διοκτικών αρχών και βέβαια και της στρατιωτική ε, πλευρά της συλλογής πληροφοριών γιατί χρειαζόμαστε και το στρατιωτικό τομέα κυρίως για ε, θέματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και συγκρούσεων. Ρωτήσατε επίσης κερδίζουμε ή χάνουμε. Μιλούμε για εγκληματική συμπεριφορά και τρομοκρατία. Ρωτήσατε εάν κερδίζουμε έδαφος, ίσως είναι καλύτερα να το πω έτσι. Εγώ θεωρώ ότι όντως κερδίζουμε έδαφος. Αργά αλλά σταθερά. Δεν είναι όμως, δεν ήρθε όμως η ώρα να επαναπαυθούμε. Είπα πριν κάτι για τις περιοχές συγκρούσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν ωστόσο να προκαλέσουν τρομοκρατική δραστηριότητα είτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε κατά συμφερόντων της Ένωσης εκτός αυτής. Μάλι είδαμε στη Γαλλία να γίνονται ορισμένες συλλήψεις ε, ε, κατά προσώπων που προέρχονται από την περιοχή αυτή του κόσμου. Αν δούμε λοιπόν τις περιοχές συγκρούσεων, αυτές οι περιοχές συγκρούσεων πάντοτε έχουν το δυναμικό να προκαλέσουν συγκρούσεις και εκτός της περιοχής τους σε βάρος οικονομικών συμφερόντων ή της ασφάλειας και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, απαγωγές στην περιοχή της Σαχάρας ε, ε, Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι μετακρατούνται όμοιροι. Αυτά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Εγώ θα ήθελα να θέσω επίσης ορισμένες ερωτήσεις, γιατί θα ήθελα να μάθω ποια εγκληματική οργάνωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα θεωρείται ως ιδεώδη εταίρο τρομοκρατών. Με την έννοια ότι έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα. Εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκρατικέ οργανώσει στην ε, Ευρώπη ε, ή στην Ιταλία ενδεχομένω. Μπορείτε να μα πείτε επίση τρομοκρατικές δραστηριότητε στις οποίες υπήρξε συνενοχή από το οργανωμένο έγκλημα. Thank you, Madam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Μακαρένκο. Απλές ερωτήσεις, ναι. Δύο απλές ερωτήσεις κάνατε, αλλά πώς να απαντήσω. Ιδεώδης εταίροι λέτε, ποια εγκληματική οργάνωση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα θα ήταν ιδεώδης εταίρος. Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι όντως έχουμε περιοριστεί λίγο στην ανατενισή μας. Όλες οι οργανώσεις εν δυνάμει νομίζω που έχουν διεθνή δίκτυα θα μπορούσαν να ε, αποτελέσουν εταίρους ε, τρομοκρατικών οργανώσεων. Η εγκληματική ομάδα ωστόσο πρέπει να διαθέτει και την βούληση να εμπλακεί σε συνεργασία με ομάδες οι οποίες εν τέλει αποσκοπούν στην αναστάτωση της ζωής της κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται η εγκληματική οργάνωση αυτά στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο ε, επιβάλλουν και τους τρόπους συνεργασίας αυτών των ε, δύο πλευρών. Αυτό που βρήκαμε εμείς είναι ότι οι παλαιά μαφία, οι παλαιές παραδοσιακές εγκληματικές οργανώσεις είτε στο Ενωμένο Βασίλειο, είτε στη Γερμανία, είτε και στην Ολλανδία. Πάντως οργανώσεις που έχουν ιστορία τείνουν να μην συνεργάζονται δεν συνεργάζονται με ε, τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι νεότερες με νεότερη ηγεσία σκέφτονται περισσότερο τι έχουμε να χάσουμε. Ας συνεργαστούμε. Και θα έχουν επομένω πρόσβαση σε δίκτυα σωματεμπόρων ή ε, δίκτυα ε, παράνομης διακίνησης όπλων. Γίνεται ένα business relationship, μια επιχειρηματική σχέση τα βλέπουμε αυτά και σαν μια κινηματογραφική ταινία. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Παύλο Εσκομπάρ να κάθεται να συμφάγει με τον Οσάμα Μπινλάδεν. Δεν ξέρω, ίσως να το κάνουν τώρα εκεί που βρίσκονται και οι δυο, αλλά ε, κάπως έτσι. Ή τέλος πάντων, μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα, γιατί τότε θα ήταν και η παρακολούθησή τους πιο εύκολη. Αλλά υπάρχουν κάποιες ε, έτσι επαφές, είναι αυτή η facilitator, που θα διευκολύνουν την μεταφορά 10 ατόμων από το Πακιστάν, για παράδειγμα, στα ευρωπαϊκά σύνορα. Α, τότε θα πούν και αυτοί, είμαστε Ισλαμιστές μαχητές και θα σας βάλουμε βόμβες. Μπορεί να είναι 10 ε, Πακιστανοί οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους ε, στη, στο Ενωμένο Βασίλειο. Θα πληρώσουμε τότε λοιπόν τους ε, ε, λαθρεμπόρους αυτούς προσώπων, πώς να πω, τους σωματεμπόρους αυτούς οι οποίοι θα τους διευκολύνουν να περάσουν και να φτάσουν στα σύνορα και να τα διαβούν εν τέλει. Τώρα, ποιος όμως παίζει ποιο ρόλο είναι ένα θέμα. Και καμιά φορά από τη δική μας την σκοπιά τα εξετάζουμε αναδρομικά. Και μετά ερχόμαστε και λέμε, «Χα, μα πώς και δεν τα είδατε αυτά τα πράγματα» Αυτά λέω και στους ε, γνωστούς μου από τις διοκτικές αρχές που έρχονται και με συμβουλεύονται. Υπάρχουν παραδείγματα που θα μπορούσα να σας πω και μάλιστα περιλαμβάνονται ορισμένα και στις εκθέσεις που έχουμε συγγραφεί. Τώρα, τρομοκρατικές δραστηριότητες οι οποίες έγιναν με συμμετοχή τρομοκρατικών οργανώσεων ε, εγκληματικών οργανώσεων μάλλον. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όπου να είπαν οι διοκτικές αρχές ότι η τάδε τρομοκρατική οργάνωση συνεργάστηκε με την τάδε εγκληματική οργάνωση για μια βομβιστική απόπειρα. Πιο πολύ πρόκειται για μια στήριξη που δίνεται μέχρι την τρομοκρατική απόπειρα. Με τις βόμβες του 2004, για παράδειγμα, είχε ε, υπάρξει συνεργασία με δίκτυα λαθρεμπορία. Τώρα αυτό το, ε, την υπόθεση στην ε, Τουλούζη, ορισμένοι είπαν ότι ήταν με το φόνο του Μύρα και των μελών τη οικογένεια του. Ο Μύρα, ωστόσο, είχε διασυνδέσεις και με, το μαχητικό, και με μαχητικούς Ισλαμιστές σε ορισμένες ομάδες, αλλά και μέσω του αδελφού του με το οργανωμένο έγκλημα. Να λοιπόν οι δύο παράλληλες αυτές πορείε ε, της ζωής ενός ατόμου, ο οποίος αντλούσε και από τι δύο αυτέ δυναμικές, ευτυχώ ή δυστυχώ τέλος πάντων, ε, αυτός ο Μοίρα θεωρήθηκε τελικά σαν μοναχικός λύκος κατά κάποιο τρόπο. Και, και, και έτσι κρίθηκε η περίπτωση αυτή. Αλλά ίσως υπάρχουν περισσότερα πράγματα που κρύβονται από πίσω. Και υπάρχουν και κάποια προφίλ άλλα, άλλων ατόμων που κρύβουν περισσότερα πράγματα γιατί οι τύποι αυτοί λειτουργούν πάνω στο όριο εγκληματικότητας, οργανωμένου εγκλήματος και ε, τρομοκρατίας. Ο άλλος που είπα πριν, ο Μουχτάτελ Μουχτάρ, είναι γνωστός στο Βόρειο Μάλι ως ο κύριος Μάρλμπορο. Ήταν επικεφαλής ολόκληρου οργανωμένου δικτύου λαθρεμπορίας τσιγάρων. Αυτή η συνενοχή δεν είναι συνοχή του είδου ε, συνενοχή μεταξύ δύο ατόμων, είναι περισσότερο συνενοχή δύο δραστηριοτήτων. Ελπίζω να μπόρεσα κάπως να σας απαντήσω. Ο κύριος Κώστερς, με ρωτήσατε αν μπορώ να σας πω μια ιδεώδη εγκληματική οργάνωση, άγνωστον, αλλά μια εγκληματική οργάνωση που θα στρεφόταν προς μια τρομοκρατική οργάνωση, θα δραστηριοποιούσε τις εγκληματικές τις δραστηριότητες, αλλά ταυτόχρονα θα συναποτελούσε μέρος τρομοκρατικής οργάνωσης. Αλλά βέβαια υπό τον πλήρη έλεγχο της τρομοκρατικής οργανώσεως. Αυτό που είναι άγνωστο σε εμάς, βέβαια, στην περίπτωση αυτή δεν μπορώ να σας δώσω με το προφίλ τέτοιας εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό θα ήταν αδύνατο να το πράξω. Για την ώρα τουλάχιστον. Επίσης, είπατε για τρομοκρατικές δραστηριότητες, τα είπε και η κυρία Μακαρένκο, όπως για παράδειγμα ε, το λαθρεμπόριο καπνού. Έχω και ένα παλαιό παράδειγμα. Στις μέρες της απαγόρευσης της κυκλοφορίας του βόηου κρέατος, με τις τρελές αγελάδες κτλ. Και βρετανικό βοδινό είχε απαγορευτεί να κυκλοφορεί. Τι έγινε λοιπόν στην δημοκρατία της Ιρλανδίας, στη Βόρεια Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδικά βόδια πέρασαν τα σύνορα προς την δημοκρατία της Ιρλανδίας και ξαφνικά έγιναν Ιρλανδικό κρέας. Να, ένα άμεσο πράγμα με όλη αυτή την ιστορία με το βόλιο κρέα. μια άμεση συνέπεια της μετακίνησης των ε, αγελάδων, των βοδιών, που ήταν απολύτως άχρηστα εκείνη την εποχή, δεν είχαν απολύτω καμιά άξια, αλλά τα πέρασαν από τα σύνορα, έγιναν, τα βαφτίσανε αυτομάτως Ιρλανδικό βοδινό και επομένως ε, οδηγήθηκαν στην κατανάλωση. Και από εκεί βέβαια βγάλανε λεφτά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μήτα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ στην αρχή, γιατί αυτή είναι η τέταρτη συνεδρίαση μου σήμερα το πρωί. Θα με ενδιαφέρε η ισορροπία στην νομοθεσία σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία. Όταν ε, είχαμε την ε, επίθεση στο Ο1. Νόμιζα ότι εδώ θα έπρεπε να δράσουμε γρήγορα, αλλά πολλές νομοθεσίες και οι ευρωπαϊκοί έχασαν το στόχο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε επικριτικοί και να μην δημιουργούμε μια κοινωνία όπου όλοι μπορεί να είναι, ο καθένας μπορεί να είναι ενδυνάμει τρομοκράτη. Και νομίζω ότι είναι λάθος που ε, η Ευρώπη προσπαθεί να βρει τρομοκράτη σε κάθε γωνιά. Και έχουμε όλες αυτές τις έρευνες, ε, τους ελέγχους στα αεροδρόμια κτλ. Όταν ε, πήγα να επισκεφθώ το Υπουργείο Εξωτερικών στην Όσικτον, μας είπαν ότι ναι, πάντοτε βρίσκουμε τρομοκράτες, αλλά Ε, όταν ρωτήσαμε συγκεκριμένα δεν θέλανε να μας απαντήσουν. Και επίσης ε, πριν κάποια χρόνια στην Ευρώπη κάποιος μας είπε αν ναι, αποφύγαμε αυτό και το άλλο. Είναι πιο γενική λοιπόν η ερώτησή μου, γιατί νομίζω ότι εδώ αφορά το θέμα της τάσης ε, που κρατά κανείς στην κοινωνία. Εγώ είμαι υπέρ του να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή εγκληματικότητας, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα. Αλλά η ερώτησή μου είναι αυτά που κάνουμε τώρα είναι ακριβή και πετυχαίνουν το στόχο ή το τίμημα είναι η προσωπική κυριότητα και ο μη σεβασμός της ιδιωτικής ζωής. Δηλαδή, σε κάθε βήμα σου στο Ηνωμένο Βασίλειο σε παρακολουθούν οι κάμερες. Ακόμη και στην κρεβατοκάμαρα γίνονται έρευνε. Δηλαδή είναι ισορροπημένη αυτή η προσέγγιση, αυτό ρωτάω. Και αν ε, λέτε ναι, βρίσκουμε όλους τους απαταιώνες, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν ε, απαταιώνες εγκληματίε, είτε είναι τρομοκράτες είτε όχι. Εγώ είμαι κάπως ε, διστακτικός για το αν κάνουμε το σωστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς οι προσκεκλημένοι μας ε, είναι ειδικοί, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Είτε μπορούν να απαντήσουν εδώ, είτε στο μέλλον. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τις ε, χρηματοοικονομικές βάσεις, ε, δηλαδή ποιοι είναι οι λογαριασμοί που στηρίζουν την τρομοκρατία. Ευχαριστώ και πάλι το λόγο έχει η κυρία Μακαρέγκο και κατόπιν ο κύριος Κώστερς. Um, Θα αρχίσω με την πιο άμεση ερώτηση για τις γραπτές απαντήσεις όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους. Ναι, σημός υπάρχει. Τώρα το πρώτο είναι μια μεγάλη συζήτηση που κρατάει για τις αντιτρομοκρατικές πολιτικές. Και σωστά λέτε ότι μετά τις 11 Σεπτεμβρίου το γεγονός αυτό καθορίζει τις πολιτικές μας. Παρόλο που ο κύριος Μπλερ ήταν πολύ πιο πίσω. Υπήρξαν όμως νομοθετικές αντιδράσεις σε αυτό. Κάποιοι μπορεί βέβαια να πούν ότι δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατόμων από τη μια και από την άλλη ο εντοπισμός των εγκληματιών και τη μορία τους. Είναι αρκετά φιλοσοφικό ζήτημα, έτσι. Οι δυτικές κοινωνίες ε, συχνά ε, λένε πρόκειται για τα δικαιώματα των ατόμων. Ωραία. Άρα αυτά πρέπει να τα προστατεύουμε. Ενώ από την άλλη μεριά οι άνθρωποι για να περάσουν τον έλεγχο στο αεροδρόμιο πρέπει να βγάλουν τα παπούτσια τους, τις ζώνες τους κτλ. Ή να εξηγήσουν γιατί αντί για 99 έχουν 100 λίρες απάνω τους κλπ. Πάντως στη συζήτηση αυτή εγώ πιστεύω ότι παραβλέπουμε τελικά παραβλέπουμε τελικά τη, τα δικαιώματα της κοινωνίας ολόκληρης Μπορεί να ε, δυσκολεύουμε λίγο κάποια άτομα, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί έτσι να σταματήσουμε μια επίθεση η οποία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάποια άτομα με τίμημα τι να το αναγκαστώ να βγάλω τις μπότες μου, τη ζώνη μου στο αεροδρόμιο. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν πόσο μακριά πάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που τέλος πάντων πιέζουμε ή παραβιάζουμε και να δούμε και από την άλλη μεριά ποιο είναι το κέρδος. Δεν πρέπει να καταλήξουμε σε μια παρανοϊκή βέβαια κατάσταση όπως είχαμε με την ΚΑΚΕΜΠΕ τη δεκαετία του 60. Πάντως, αν πιστεύουμε ότι αν κάποιος πιστεύει ότι εγώ είμαι εμπλεγμένο σε εγκληματικές δραστηριότητε και γι' αυτό θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνομιλία μου με τη μαμά μου ή με δεν ξέρω εγώ τι ή να βάλουν κάμερες εκεί που βγάζω βόλτα το σκύλο μου για να είναι σίγουροι ότι δεν συμβαίνει τίποτα το περίεργο, ε, ας είναι αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα ατομικά δικαιώματα, τα άτομα του ατόμου είναι η προτεραιότητα. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι φιλοσοφική ερώτηση και φιλοσοφική και απάντηση. Τι θέλουμε να διασφαλίσουμε, τι θέλουμε να προστατεύσουμε. Ανάλογα με αυτό έρχεται και απάντηση. Ευχαριστώ, κύριος Κώστερ. Αν υπάρχει ισορροπημένη προσέγγιση ήταν η πρώτη ερώτηση. Για μας, με κάθε σεβασμό, είμαστε υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου. Οπότε, τι κάνουμε, προστατεύουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό σημαίνει και τα ατομικά τους δικαιώματα. Οπότε, ακολουθούμε την υπάρχουσα νομοθεσία η οποία μας επιτρέπει να επιβάλλουμε τον νόμο ως έχει. Είναι περισσότερο δηλαδή θέμα πολιτικής ε, δύναμης παρά θέμα ικανότητας επιβολής του νόμου από τους ε, αξιωματούχους, αστυνομία κλπ. Κατά πόσο το τίμημα είναι υψηλό. Και πάλι για μένα είναι πολιτικό το ζήτημα. Ρωτήσατε επίσης, υπάρχει καμιά γραπτή έκθεση για την χρηματοδότηση του κλίματος. Ναι, η Europol, επειδή ο κύριος Κίρχοφερ της το ζήτησε, ετοίμασε μια τέτοια έκθεση που είναι του Μαΐου του 2012. Παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον κύριο Κίρκοβερ στο Συμβούλιο του 2012. Ευχαριστούμε κύριε Κώστερς. Παρακαλώ, Μπιλ. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Κώστερς μόλις τώρα για τον αντιτρομοκρατικό συντονιστή στην Ένωση. Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι ως ενεργεία αστυνομικός δεν θέλετε να συζητήσετε για ε, ε, θέματα πολιτικά. Έχουμε όμως έναν παλαιό Ολλανδό ε, φιλελεύθερο, τον κύριο Ντεφρίς, ο οποίος έγινε συντονιστής αντιτρομοκρατικών ενεργειών της Ένωσης και μετά παρετήθηκε διότι μου παραπονέθηκε εμένα και ελπίζω να μην έχει αντιρρήσει να το πω, ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Γι' αυτό και σε ξανακάνω το φιλοσοφικό ερώτημα, τα πάμε καλύτερα ή εξακολουθείτε να αισθάνεστε μια πλήρη απογοήτευση. Για να είμαι ειλικρινή, κάθε συζήτηση για τον αντιτρομοκρατικό συντονιστή, κοιτάξτε, μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο. Συντονίζει ή προσπαθεί να συντονίσει τι προσπάθειε των κρατών μελών ο άνθρωπο αυτό. Και είμαστε σε συνεχή επαφή με τον κύριο Ντεκερκόφε. Και από τότε που ξεκίνησε ο κύριος Δευρή ε, και από τότε που τον αντικατέστησε ο κ. Δικερκόπε, είχαμε κάποια επιτεύγματα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλά επιτεύγματα στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι εδώ την καθημερινή δουλειά μου, Εργάζομαι τώρα για την Europol από το 2008 και πάλι βλέπω αύξηση στην οργανωτικότητά μας. Βλέπω ότι υπάρχει αύξηση στις πληροφορίες που μας στέλνονται. Βλέπω αύξηση στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών στο να παρουσιάσουν συγκεκριμένα προγράμματα, Παίρνουμε το σχάρι, έχουμε το σχέδιο δράση για τη ριζοσπαστικοποίηση, για τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, για την ασφάλεια των εκρηκτικών και όλα αυτά τα σχέδια δράση για μα έχουν αποτέλεσμα. Γιατί σε αυτά τα σχέδια δράση ε, βλέπουμε δραστηριότητε ε, να πηγάζουν. Αν δείτε το σχέδιο για την ασφάλεια των εκρηκτικών, ε, τώρα υπάρχει ένα σύστημα που λειτουργεί ε, και παραδείγματος χάρη μας βοήθησε πάρα πολύ στην τελευταία επίθεση στην ε, Βουλγαρία, στον Μπουρκάς. Ε, έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι το έργο του αντιτρομοκρατικού συντονιστή να μας διαχειρίζεται όλους ως ομάδα είναι ένα δύσκολο καθήκον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κώστερς. σε σχέση με την επίθεση στη Βουλγαρία την περασμένη εβδομάδα μία αντιπροσωπεία α, της ΚΡΙΜ και της ΛΥΜΠΕ αλλά και ε, ο διευθυντής της Ιεροπόλη μας ε, μίλησε για το πώς μπόρεσαν ε, οι αξιωματικοί της ε, Europol ε, να φτάσουν και επί και ότι ε, οι δικοί σας αστυνομικοί κατάλαβαν αμέσω ότι υπήρξε εμπλοκή κάποιων λιβανέζικων πυρήνων γιατί βρήκαν εκεί κάποια εργαλεία που είχαν χρησιμοποιηθεί για να φτιαχθεί η βόμβα έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και μια δραστηριότητα πληροφοριών πέρα από το συντονισμό που είναι πάρα πολύ καθοριστική. Άλλες ερωτήσεις? Όχι. Ευχαριστώ λοιπόν τους ε, ομιλητές. Θα διακόψουμε μέχρι το απόγευμα. Θα ξαναρχίσουμε στις 3.